Good afternoon. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. May I ask you to take your seat? Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε για να αρχίσει η συνεδρίαση. I'm sure we'll see more colleagues coming. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι αργότερα. Ε, για μια ελπίδα ζούμε. Yes, yes, these are troubles in flying and traveling in a way. Ξέρω, το ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τις πτήσεις, χειμωνιάτικα, Δευτέρα, είναι όλα αυτά προβληματικά. Εν πάση περιπτώσει, σας καλωσορίζω όλους τους παρόντες και θα περιμένουμε και τους υπολείπους συναδέλφους. Κυρίσω την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι η ε, τακτική μας συνεδρίαση. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Έχετε λάβει το σχέδιο μερίσια διάταξη. Έτσι δεν είναι στα χαρτιά σας. Θα σας πρότεινα μια μικρή αλλαγή στο σχέδιο μερίσια διάταξη. Νομίζω έχετε λάβει γνώση, σας ειδοποίησε την Παρασκευή Γραμματεία, αλλά στο επαναλάβω για καλό και για κακό. Η κυρία Γιώτοβα έχει σημαντική ανελημμένη υποχρέωση στη Βουλγαρία και κολλείεται να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Γι' αυτό θα σας πρότεινα το σημείο 3 να αφαιρεθεί ε, από την ημερήσια διάταξη τη σημερινή και να μπει αύριο το πρωί στις 9. Και να αλλάξει με το σημείο του κυρίου Τόμασιτ σε επαριθμών 8. Και επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω την κυρία, συγγνώμη, Τόμασιτς, ε, που ε, δέχτηκε να κάνει αυτή την αλλαγή με την κυρία Γιώτοβα. Αν συμφωνείτε λοιπόν θα δούμε σήμερα την έκθεση της κυρίας Τόμασιτς και αύριο της κυρίας Γιώτοβα. Συμφωνείτε, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με αυτή την αλλαγή και προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Έμαθα ότι κάποιοι συνάδελφοι ε, είχαν διάφορα προβλήματα και ανελημμένες υποχρεώσεις και απουσιάζουν η κυρία Μάλκοβα, η κυρία Νταντσίλα και μερικοί εισηγητές, τουλάχιστον δύο, η κυρία Μάλετιτς και δύο εισηγητές, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Το εξήγησα στην κυρία Νταμάτο, ζητώ συγγνώμη κύριε Βανίστεροι. Έχουμε όμως συναδέλφους που θα κάνουν τις παρουσιάσεις των θεμάτων τους Η θα μπορέσουμε να καλύψουμε την ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη μου ανακοίνωση αφορά την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών στο Λουξεμβούργο 26 και 27 Νοεμβρίου κατόπιν ε, προσκλήσεως της ε, Λουξεμβουριανής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άτυπες συνεδριάσεις των ε, αρμοδίων ε, Υπουργών για την Αστική ε, Πολιτική και την Εδαφική Συνεργασία έλαβαν χώρε 26 και 27 του μηνό, την περασμένη λοιπόν Πέμπτη και Παρασκευή. Ε, μαζί με τον κύριο Ομαρζέ προσωπήσαμε την Επιτροπή μας και συζητήσαμε την πρόοδο στην εδαφική συνοχή, διάφορα εδαφικά σενάρια και οράματα και σκέψεις για διασυνοριακή συνεργασία, θεματολόγιο, προκλήσεις της πόλης από την κατάσταση των προσφύγων. Το σχέδιο συμπερασμάτων εγκρίθηκε από όλα τα μέλη του Άτυπου Συμβουλίου. Γενικά η συζήτηση δεν ήταν επίμαχη, δεν ήταν σύγκρουσιακή. Για το θέμα των προσφύγων και την κατάσταση της πόλης έγιναν διάφορες προτάσεις και μπορώ να πω ότι η άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών έχει παρεμφερεί η μερίσια διάταξη με τη δική μας. Μας απασχολούν τα ίδια θέματα. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω όλους τους Υπουργούς για τις ε, εκθέσεις που συζητούμε και τις ε, επερχόμενες εκθέσεις και εκείνοι με ενδιαφέρον άκουσαν και κατάλαβαν ότι εργαζόμαστε με την ίδια ταχύτητα για τα ίδια θέματα, παράλληλα με το Συμβούλιο δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Αλλιώς μπορώ να σας τα πω και διμερός και πιο άτυπα να σας εκθέσω τις απόψεις μου και τις εντυπώσεις μου από το Υπουργικό αυτό Συμβούλιο το άτυπο. Τελευταία ανακοίνωση θα ήθελα να σας θυμίσω, με χαρά το κάνω, ότι ε, σας προσκαλούμε σε μια δεξίωση στις 6.30 απόψε στο Γεχούντι Μενουχίν στο διπλανό κτίριο, PHS. Ε, δεν είναι ακριβώς χριστουγεννιάτικο αυτό, αλλά είναι μια αποχαιρετιστήρια για φέτος εκδήλωση, αφού είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος. Καλή ευκαιρία. Λοιπόν, για να τα πούμε σε ένα πιο άτυπο και πιο χαλαρό περιβάλλον και να ανταλλάξουμε ευχές για τα Χριστούγεννα και το Δεκέμβριο φυσικά πριν φτάσουμε στα Χριστούγεννα, να έχουμε επιτυχίες στις εργασίες μας. Αυτά από ανακοινώσει και θα περάσουμε μέσω στο τρίτο σημείο πρώην 8. νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξη στην πολιτική συνοχής 2014-2020. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση και τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Η συγκήτρια είναι η κυρία Τόμασιτς. Σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης στην πραγματικη περιοδο περίοδο 2014-2020 έχουμε δύο νέα εργαλεία για την εδαφική συνοχή και να επιτευχθούν οι στόχοι και αυτά είναι αυτά που σας προανέφερα, το ITI και το CLLD. Αφορούν όλα τα ταμεία που καλύπτονται από του αντίστοιχους κανονισμούς. Αποφασίσαμε να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλίες πρωτοβουλίας για τα δύο αυτά νέα μέσα και η συγγήτριά μας Τον Οκτώβριο ήδη μας παρουσίασε την έκθεση, τις πρώτες απόψεις. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Προτείνω προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, για να ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας στις 15 και 16 Φεβρουαρίου του 2016. Ορισμένοι σκιώδεις παρευρίσκονται, άλλοι πάλι όχι. αλλά τους εκπροσωπούν άλλοι συνάδελφοί τους. Έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μέρια Χαπάκα, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα δώσω μέσα το λόγο στην εισηγήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδους, ε, συζητητές για τις προτάσεις και τη συνεργασία τους ε, που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Αυτή η έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας εστιάζεται σε κάποιες πρώτες εμπειρίες και στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση των νέων εργαλείων εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής ε, 2014-2020. Παρέχει επίσης μια ανάλυση των εμποδίων ε, για την υλοποίηση και συστάσεις για τη μελλοντική υλοποίηση για τα κρατη μελικίνα που δεν ε, τα είχαν οθετήσει πλήρω ε, στο χρονικό διάστημα 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιαστεί περισσότερο στην εδαφική συνοχή εντός του νομοθετικού πλαισίου για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η περίοδος 2014-2020 περιλαμβάνει προβλέψεις για ειδικά εδαφικά μέσα, το CLLD και το ITI, που θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει πολλές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση ώστε να εξευρεθούν ε, αποτελεσματικές λύσεις. Απαιτείται ε, ε, μια προσέγγιση που να μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες περιοχές και στα χαρακτηριστικά τους. Η προσέγγιση αυτή θα απαιτήσει ισχυρότερη δεσμεύση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης ώστε να επιτευχθεί συνεργασία και να συντονιστούν οι δραστηριότητες ε, για την επιδεύξη των κοινωνικών στόχων. Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, η υποχρεωτική αστική διάσταση χρησιμοποιείται για τις ε, δράσεις αηφορού ανάπτυξης. Ένας από τους τρόπους εκπλήρωση αυτού του κριτηρίου είναι μέσω της ε, ITI, τη ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση, η οποία καθιστά δυνατό για τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα ταυτόχρονα, αντλώντα ε, κονδύλια από πολλαπλού άξονε προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν την υλοποίηση μια ε, ολοκληρωμένη στρατηγική για μια συγκεκριμένη περιοχή. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ενσωματώσει τα CLLD στι ε, συμφωνίε εταιρικέ σχέσει του το οποίο δείχνει πόση σπουδαιότητα έχει η τοπική ανάπτυξη τη σημερινή μέρα. Ε, το κλειδί για μια επιτυχή ε, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω είναι η κατάλληλη κατανομή ευθυνών και χώρις ευθυνών σε τοπικούς ενδιαφερόμενους και η υλοποίηση τοπικών περιφερειακών στρατηγικών. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν ιδιαίτερα την υιοθέτηση μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω ούτε να εκχωρήσουν ε, ευθύνες σε τοπικές ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σημαντική ανάπτυξη μια στρατηγική που θα ενημερώνει και θα παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στους ενδιαφερομένους, ειδικότερα στους δημόσιους οργανισμούς που χρειάζεται τεχνική και οικονομική υποστήριξη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα στα πρώτα στάδια της υλοποίησης. Το ζήτημα της ανάληψης ευθύνης ε, για την επίτευξη αποτελεσμάτων από τοπικές ομάδες είναι κέρια σημασία για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα των αναπτυξιακών στρατηγικών. Για να επιτύχει το εργαλείο αυτό πρέπει να υποστήριζεται από όλα τα πολιτικά επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Γι' αυτό το λόγο κάνω έκκληση προς την Κομισιόν ε, να ε, χρησιμοποιήσει τι εξουσίε τη και να εκδώσει συστάσει προ τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνηση για την υλοποίηση του CLLD και του ITI. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις για την υλοποίηση του ITI, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι τοπικοί εταίροι θα πρέπει να παίζουν ρόλο κλειδί στην υλοποίηση τη στρατηγική. Θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο στις ευθύνε που σχετίζονται με τη διαχείριση, την παρακολουθήση και τον έλεγχο. Επίσης καλωσορίζω και την συμμετοχή διαφόρων εταίρων από τοπικέ ε, ομάδε δράσης. Ωστόσο, ο κανόνας ότι οι δημόσιες αρχές ε, δεν πρέπει να έχουν ε, δικαιώματα ψηφοφορία πάνω από 49% σε, ε, τοπικές ομάδες, σε ομάδες τοπικές δράσης μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση του CLLD λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης στις ενδιαφερομένες ομάδες. Έτσι λοιπόν κάνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί προσεκτικά τους κανόνες και την υλοποίησή τους ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές όπου μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα αυτές οι απαιτήσει και να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκδώσει συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Είναι πολύ σημαντικό να εμπλακούν οι νέοι στην υλοποίηση της CLLD. Οι νέοι συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο λόγο και συχνά ε, χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητοι ε, μεγάλο ποσοστό νέων δεν έχει πρόσβαση σε ε, εκπαίδευση, σε κατάρτιση, σε επαγγελματική κατάρτιση ε, και ταυτόχρονα τα ποσοστά ενεργείας ε, των νέων υπερβαίνουν το 50% σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η συμμετοχή λοιπόν των νέων στην CLLD μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό πολύ αποτελεσματικότερα. Επίσης θα ήθελα να κάνω και έκκληση προς τα κράτη-μέλη να παράσχουν επιπλέον υποστήριξη και συμβουλές σε δήμους ε, μικρούς ε, και σε μικρές περιφέρειες που συχνά έχουν ελάχιστους πόρους ε, και ελάχιστες δυνατότητες και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του διοικητικού βάρους. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο του CLD και του ITI πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες απλούστευσης του πλαισίου ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των εργαλείων αυτών με αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό τον λόγο καλωσορίζω τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου ανεξάρτητων ε, ειδικών που θα παρακολουθούν τη διαδικασία απλούστευσης προ όφελο των δικαιούχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Επίση, καλωσορίζω το έργο της Κομισιόν στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας του Better Regulation. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε ε, όσον αφορά την εκπόνηση των συστάσεων, διότι απλούστευσε ένα κράτος μέλος μπορεί να σημαίνει ε, πιο περίπλοκες διαδικασίες ένα άλλο. Ε, θέλω λοιπόν να παροτρύνω την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν, να προλιάνουν το έδαφος για να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ διοικητικών αρχών και στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων επίσης θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή ενημέρωση προς τους πιθανούς δικαιούχους ώστε να μπορούν να ε, αμφισβητήσουν ε, τυχόν διοικητικέ αποφάσει. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο ε, συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και κομισιών όσον αφορά τι κατευθύνε γραμμέ. Οι κατευθύνε γραμμέ πρέπει να εκπονούνται παράλληλα με τι νέε νομοθετικέ προτάσει στον τομέα τη πολιτική συνοχή και μετά να ακολουθούν περαιτέρω επικαιροποιήσει σε περίπτωση αλλαγών στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα δώσει σε όλου τη δυνατότητα να υποβάλουν τα έγγραφα για τις κατευθυντήρες γραμμές έγκαιρα και κατά τις ε, διαπραγματεύσεις μπορούν να παρέχονται περισσότερες συμβουλές. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και συστάσεις και προσλέπω στη συνεργασία μας. Πιστεύω ότι η κοινή μας προσπάθεια θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καλό σχέδιο κειμένου το οποίο θα υιοθετηθεί ε, εύκολα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. από τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Βάνα. Uh, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτη μου δίνετε το λόγο με τη σειρά, είναι κάπως ασυνήθιστο. Ο συνάδελφος Κρέλιτς των Πρασίνων είναι σκιώδης ηγητής. Θα ήθελα ε, να ζητήσω συγγνώμη ε, για την απουσία του. Έχει ανελημμένες πολιτικές υποχρεώσεις στην Κροατία και ε, θα θέλαμε να μοιραστούμε τις εξή απόψεις μαζί σας. Ευχαριστούμε την κυρία Τόμασιτς πάρα πολύ για το σχέδιο έκθεσής της και καλωσορίζουμε την ανάγκη για ένα νέα, έκθεση πρωτοβουλίας μάλλον για τα νέα εργαλεία. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ε, συμμετέχει ε, και παντού, όχι μόνο στην ανάπτυξη της υπέθρου. Χρειάζεται πλέον εκχώρηση ε, ε, αρμοδιοτήτων, αλλά υπάρχουν ακόμα ισχυρές αντιστάσεις από διοικητικούς και πολιτικούς φορείς και καλό θα ήταν αυτές να καμφθούν έτσι ώστε οι λύσεις να είναι βιώσιμες. Το CLLD δεν είναι ένα ε, απλό έργο διαχείρισης και άσκησης πολιτικής από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να συμμετέχουν ε, όλοι οι ντόπιοι ε, εμπειρογνώμονες να αξιοποιούνται και έτσι δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας για την ευφυή ε, ειδίκευση, πράγμα που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη παντού, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη σημασία και τα πλεονεκτήματα από τα νέα έργα. Η υποστήριξη και η ενίσχυση του τοπικού επίπεδου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως ομάδα και πιστεύουμε πολύ ότι η κυρία Τόμασιτς θα υποστηρίξει τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And, uh, Ευχαριστώ. Mr. Santos. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, ο κύριος Σάντος, που μιλάει ξανά όμως ο κύριος Ροντρίγκες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Η Ελιάνε Ροντρίγκες ε, δυστυχώς δεν ε, μπορούσε να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω και να παρουσιάσω τη θέση της επειδή είναι σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστή την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έχει κάνει. Ο στόχος είναι να δοθεί η αξία που αναλογεί στις περιοχές, αυξάνοντας το δυναμικό τους και μέσα από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη να μειώσει την ασύμμετρη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που οδηγεί σε αποδυνάμωση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα που κατοχυρώνεται όμως από τις συνθήκες Λισαβόνας, έτσι και την οικονομική οικονομική και κοινωνική συνοχή, διότι είναι θεμελιώδη στόχος μιας Ευρώπης που είναι όλο ένα και εγκύτερη στου πολίτες της. χάρη στην συνεργασία λοιπόν μέσα από αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε πάρα πολλά ωφέλη βελτιστοποιώντας και εξορθολογίζοντας μια κρίσιμη μάζα η οποία ε, εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των πόρων ως προς την προώθηση ε, προγραμμάτων ε, συνεργασίας διαφόρων περιοχών, τονίζοντας έτσι την περιφερειακή και τοπική διάσταση αλλά και τη συνεργασία που μπορεί να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο. Ε, θα πρέπει λοιπόν, ε, χρησιμοποιώντας αυτούς τους δύο διαφορετικούς μηχανισμούς επενδύσεων, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες, διότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση για τα προγράμματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ίδιες οι περιοχές συμμετέχουν στην κατάρτιση και στην υλοποίηση των προγραμμάτων μέσα από νέες εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εξασφαλίζοντας σε μια αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και επίσης εξασφαλίζοντας και μια ισορροπία ως προς τις υλοποιηθήσεις επενδύσεις. Ε, αυτές οι συμφωνίες εταιρικέ σχέσεις ε, θα διευκρινίζουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες ε, των συμβαλωμένων μερών πρέπει να οριστούν επακριβώς για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αυτές οι αρμοδιότητες σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Λογική απόρρια αυτού του επιχειρήματο είναι είναι ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ε, ε, υλοποιήσουν το δικό τους ρόλο. Είναι περίπλοκοι οι νέοι μηχανισμοί και γι' αυτό χρειαζόμαστε ειδική κατάρτιση για το προσωπικό των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ε, χρειάζεται ενημέρωση και κατάρτιση η οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οδηγώντας μας έτσι σε μια προσέγγιση πολυταμιακή. Ε, έτσι με τις νέες αυτές δομές ενισχύεται η τοπική και περιφερειακή διάσταση ούτως ώστε να επιτευχθεί μέχρι στη δυνατή ευρωπαϊκή συνεργασία. Χρειάζεται ευελιξία στους κανόνες και αυτό θα εξασφαλιστεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ξεκάθαρων κανόνων, ώστε να ε, μειώσουμε τι ανισότητε ανάμεσα στι περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνε θα πρέπει να είναι ομοιόμορφοι σε όλε τι περιοχέ και δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στο αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε τι ε, ε, δυσκολίε που μπορούν να ανακύψουν και όχι να προσπαθήσουμε να τι διορθώσουμε μόλι συμβούν. Και κυρίω αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι ως προς το τελικό προϊόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν σε συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να φροντίσει για την ενημέρωση σε σχέση με το νέο σύστημα ε, και ε, να παράσχει τα απαιτούμενα κίνητρα στις περιοχές, σε επιμένους περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουν ποιο θεμελιώδη ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν για να ε, τελεσφορήσει η νέα πολιτική συνοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η παρέμβαση που μου ζήτησε η Ελιάνα Ροντρίκης να σας παρουσιάσω. Thank you very much, Mr. Van... Ευχαριστούμε πολύ, ο κ. Βανίστελρο. Um, Ευχαριστώ. Ε, ο σκιώδης εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ο κύριος ε, Μπούντα. Ε, είναι παρόν, είναι στο δρόμο. Καλά, να πω εγώ τα δικά μου σχόλια τότε. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση. Είναι γεγονός αυτό. Βραχυπρόθεσμα περιμένω και θέλω να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται ε, για την έκθεση για το άρθρο 16 σημείο 3 για την ανάλυση ε, στο περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ε, συμβολέων των εταιρικών για να δούμε στην ουσία τι γίνεται. Ρώτησα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πόσα λεφτά μιλάμε γιατί ε, είναι αυτό το εργαλείο εθελοντικό, είναι προαιρετικό. Γίνονται συμφωνίες. Για ποια ποσά μιλάμε λοιπόν, για ποσοστά αν θέλετε, αν δεν έχετε ποσά, ε, του πλαισίου που έχουμε για τις επενδύσεις στα ΕΣΠΑ, στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, και η δεύτερη ερώτηση, θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά πράγματα για το μέσο αυτό. Ποια είναι ε, οι δυσκολίες και οι περιορισμοί. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε κονδύλια για ενοποιημένη χρήση, ο κόσμος αρχίζει να φοβάται. Ε, όχι στην αρχή, αλλά στο τέλος, όταν κλείνουν οι λογαριασμοί. Και αρχίζουν όλοι οι δικαιούχοι ε, να αγωνιούν ε, ότι δεν έχουν ε, τηρήσει όλους τους κανόνες. Άλλους κανόνες έχει το κοινωνικό ταμείο, άλλο το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, οπότε αυτό θα πρέπει να το χειρίζονται οι αρμόδιοι, αλλά ποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς λειτουργεί αυτό, θα μπορούσε να μας απαντήσει λίγο περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τα άλλα, η έκθεση επαναλαμβάνω είναι πολύ επίκαιρη, κανονικά θα έπρεπε να είναι μια έκθεση εφαρμοστική. Γιατί κοιτάμε πώς έχει στην πράξη εφαρμογή αυτών των θεμάτων και τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, τώρα προ το παρόν είναι ευκολόγια και θα είναι στα χέρια των ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθούν την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων. Αυτά είναι τα βασικά μου προβλήματα ή προβληματισμοί και ερωτήσεις και τα σχόλιά μου υπογραμμίζω πάρα πολύ ότι είναι στην καλή κατεύθυνση φυσικά για τους κανονισμούς που έχουμε αυτή την περίοδο. Κάτι που εκκρεμεί λίγο είναι έχουμε μπει στην ουσία. Είναι μια δυνατότητα, είναι ένα πυροτέχνημα, είναι ένα ε, τέχνασμα. Έχουν συμφωνίες για θεματικές ε, ε, συγκεντρώσεις, για μια συντονισμένη προσπάθεια ή όπως έχουμε δει στο παρελθόν το Leader και άλλα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, για τα χωριά, τις σημειαστικές περιοχές και τις αστικές περιοχές θα γίνει ουσιαστική δουλειά ή απλώς εκεί πέρα σηκώνουμε κονιαχτό για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Ε, πού είναι το, το κέντρο βάρους και ισορροπία. Κατά ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να μιλήσω εκ μέρου του σκιώδηση γιατί του κ. Ιακωτσίτς ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ ειλικρινά την κυρία Τόμασετς. Ε, το σχέδιο εκθεσ αυτό είναι ιδιαίτερα πλήρες. Ωστόσο, έχω κάποια επιπλέον σημεία που θα ήθελα να θίξω. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, bottom-up, όταν αναφερόμαστε σε τοπική κοινωνική εδαφική ανάπτυξη. Πρέπει να υπογραμμιστεί, να λοιπόν αυτή η διάσταση, η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω από εμάς ως Επιτροπή Ρέτζι για τη διαχείριση των κονδυλίων και εκεί έχω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, βάσει κάποιων ε, ποσών που είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ελάχιστες χώρες έχουν επιλέξει πραγματικά πολυταμιακή προσέγγιση. Και αυτό είναι περίεργο, διότι αυτός ήταν αρχικά ο σκοπός του ITI ε, και της ε, προσέγγισης ε, της ανάπτυξης που κατευθύνεται από τις τοπικές κοινότητες. Φυσικά η πολυταμιακή προσέγγιση θεωρητικά είναι εφικτή, αλλά αν δούμε πώς γίνονται πραγματικά οι συνέργειες στην πρακτική, ε, όσον αφορά λοιπόν την υλοποίηση, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητε είναι περιορισμένε. Οι πραγματικέ συνέργειε επιτυγχάνονται πραγματικά όταν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν και άλλα ταμεία. Όχι μόνο το, ε, ε τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο ή το ERDF. Δεν ξέρω, ίσω θα μπορούσε να το απαντήσει η εισηγήτρια. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολυπλοκότητα των κανονισμών, αν είναι θέμα διοικητικού φόρτου. Αν αυτές είναι οι αιτίες ε, που εμποδίζουν ε, την εφαρμογή της πολυταμιακής προσέγγισης ενδεχομένως να είναι η έλλειψη βούλησης ε, σε κεντρικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Η δεύτερη μου παρατηρήση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και τους Δήμους ε, με ε, έγγραφα με κατευθυντήρες οδηγίες ε, για το άρθρο 7, για άλλε προσεγγίσει, αλλά για το ITI η Κομισιόν έχει εκδώσει μόνο κάποια σενάρια. Ήθελα να δώσει καλύτερε κατευθυντήρε γραμμέ η Κομισιόν, ε, ώστε να καθοδηγήσει τι ε, περιφέρειες και του Δήμου που θα επιθυμούσαν να αναπτύξουν τέτοιου είδου προσεγγίσει από κάτω προ τα πάνω. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να εκδώσει καλύτερα έγγραφα ε, ιδιαίτερα εν ώψη των συζητήσεων για τη νέα νομοθεσία μετά από, την, από το 2020. Μεταδείχνει τη διάκριση μεταξύ της κρίσης των ITI για αστικές περιοχές, ε, για δήμους ε, και εκτός δήμων. Το αστικό θεματολόγιο, αυτό που γίνεται στους δήμους, πρέπει φυσικά ε, εκεί να εστιάζουμε, να τονίζουμε την προσέγγιση ATI. Ε, ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν υλοποίηση και συμφωνώ με τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Το, η έκθεση, αυτή είναι έκθεση υλοποίηση περισσότερο. Πρέπει να εστιαστούμε στο πώ γίνονται πρακτικά τα πράγματα, πώ μεταφράζουμε τη θεωρία σε πρακτική και να εκδώσουμε συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο που θα ήθελα να θίξω με ανησυχεί όταν συζητάμε για αποτελέσματα ε, που θα αποδώσει η ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Κατά την άποψή μου, μικροί οργανισμοί θα χαθούν μέσα στην πολυπλοκότητα των κανονισμών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, όταν μιλάμε για εδαφική ε, ανάπτυξη, να έχουμε και επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Ε, γι' αυτό μιλάμε για προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Γι' αυτό θα ήθελα τα κράτη-μέλη να υπογραμμίσουν την σπουδαιότητα των πρωτοβουλίων CRLD και να παρέχουν και στους τοπικούς παράγοντες αλλά και στα κράτη-μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τα εθνικά πλαίσια πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναι, σας είδα κύριε Μπούντα διότι ο κ. Βανίστελ Ρόι μόλις παρουσίασε αυτό που είχατε να πει εκ μέρους σας κάποια πράγματα. Φυσικά θα σας δώσω το λόγο αλλά να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Νταμάτο για να κλείσουμε τον κύκλο που ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους που ήθελαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και μετά θα σας δώσω το λόγο κύριε Κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι η ανάλυση των ωφελών και των επικρίσεων για αυτά τα δύο μέσα είναι απολύτως απαραίτητη για το διάστημα 2014-2020, ειδικότερα σε αυτή τη φάση από τις πληροφορίες που έχουμε από την Κομισιόν. Τα μέσα αυτά, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, θα προσθέσουν αξία στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Μπορούμε να πούμε ότι ε, για κάποια θέματα αποτελούν χάρτη καθοδήγησης ε, για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ διαφόρων διοικητικών και εδαφικών επιπέδων που συμμετέχουν στο νέο προγραμματισμό πολιτικής συνοχής. Για να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα είναι σημαντικό να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες περιγράφονται πολύ καλά στο σχέδιο κειμένου του συναδέλφου. Αυτό που μου φαίνεται ε, ότι ξεχωρίζει είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των περιφερειακών και των εθνικών αρχών και των τοπικών αρχών. Ε, τα κράτη-μέλη διστάζουν να υιοθετήσουν την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Όλοι συμφωνούμε για αυτό το επιχείρημα. Αυτή η προσέγγιση όμως θα βοηθούσε μέγιστη συμμετοχή των υποπεριφερειακών παραγόντων ε, βάσει των ικανοτήτων τους και των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Δεν οφείλει όμως να το αρνηθούμε, αυτή ο δισταγμός οφείλεται σε κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες του περιφερειακού και του τοπικού επίπεδου. Σε αυτά τα επίπεδα λοιπόν πρέπει να παρασχεθεί επαρκής τεχνική αρρώγη, δηλαδή κάποια συνοδευτική βοήθεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη κάνει εξαιρετικό έργο συντονισμού με την ομάδα ειδικών για την πολιτική συνοχή και τα αστικά θέματα. Ωστόσο, σκόπιμο θα ήταν να γίνεται και προπαρασκευαστική εργασία και κατά την φάση ε, εκπόνησης του προγραμματισμού. Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχική τοπική ανάπτυξη ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ τοπικών ομάδων και στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης δημόσιου ε, και ιδιωτικών ε, οργανισμών εξισορροπώντας την αποτελεσματικότητα του μέσου, την απλούστευση και την απαραίτητη διαφάνεια. Για να ολοκληρώσω, η πρόταση της συγγήτριας με την οποία αναλύει κατά πόσο στην επόμενο προγραμματισμό μπορεί να προταθεί η υποχρεωτική ποσόστοση για τις συμφωνίες εταιρικής σχέση σε κάθε κράτος μέλος, αντί να είναι προαιρετική, τα κράτη-μέλη, αφού θα δουν τα αποτελέσματα, πιστεύω θα πρέπει να προβούν σε κάποια ανάλυση των επιδόσεων, όχι μόνο των ε, ποσών που δαπανήθηκαν. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν προσεκτικά να δούμε τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ. κυρία Μπρέσο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα μέσα αυτά, όπως υπόθηκε μόλις, ε, ουσιαστικά υπάρχουν εδώ και καιρό. Η καινοτομία της, του τρέχοντος προγραμματισμού είναι η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών ταμείων όπου ξαφνικά διασταυρώνονται με περίπλοκο τρόπο μέσα τα οποία ήταν ήδη από μόνο τους περίπλοκα διότι σχετίζονταν με θέματα τοπικής ανάπτυξης ε, δηλαδή ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, όχι μόνο θεματικά. Ε, και αυτό περιπλέκεται με την έννοια της χρήση των πολλαπλών ταμείων, το οποίο περιπλέκει περισσότερα τα πράγματα λόγω των πολλαπλών κανονισμών, μέσω των οποίων δημιουργούνται πολλές δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπογραμμίσουμε αφενός τη σπουδαιότητα αυτών των μέσων για να συμμετέχουν πλήρως ε, οι Δήμοι στις ε, αναπτυξιακές πολιτικές. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα είναι ε, κέρια σημασίας διότι αυτά είναι κλασικά τα καταλληλότερα ε, προγράμματα για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Αν θέλουμε για να συμμετέχουν και οι μικρότεροι οργανισμοί, κομοπόλεις, αστικές, αστικές αγροτικές περιοχές, μικρές αστικές περιοχές, εκεί ίσως ε, να είναι καταλληλότερη η χρήση των CLLD. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι δυνατή η χρήση των πολλών ταμείων. Διότι πολύ συχνά το πρόβλημα ήταν πιο ότι ο προγραμματισμός που γινόταν σε ε, τοπικό επίπεδο, αυτός ο προγραμματισμός bottom-up, ε, στον οποίο αναφέρθηκαν όλοι, ε, προσέκρουε σε ένα θέμα, στο θέμα ότι δεν ήταν δυνατή η χρηματοδότηση ορισμένων ε, τομέων ε, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου που είχε επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει η Κομισιόν να εξηγήσει καλύτερα το πλαίσιο στο οποίο μπορούν, το οποίο διέπει τη χρήση των πολλών των ε, ταμείων. Κάτι που δημιουργεί πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες για τους ανθρώπους που προγραμματίζουν τέτοια προγράμματα. Διότι πρέπει να διαβάσουν πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς και τα πράγματα περιπλέκονται ιδιαίτερως. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να επανεξετάσει αυτά τα δύο ε, μέσα Εξαιρετική σπουδαιότητα για την ολοκληρωμένη ε, τοπική ανάπτυξη, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να παρεμποδιστούν από την εφαρμογή της πολυταμιακής προσέγγισης, η οποία ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεύτερον, ε, πιστεύω, και θα συναντηθούμε και με την ε, κυρία Επίτροπο για θέματα πλούστευσης για όλα αυτά τα μέσα απαιτείται απλούστευση, θα μπορούσε να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, για, κυρίως γιατί πρόκειται για μια σειρά πολύ μικρών δράσεων. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν ε, ο έλεγχος ε, να εφαρμόστε στο συνολικό αποτέλεσμα θίγοντας τα ζητήματα των ε, ε, μικρών ελέγχων ε, σε επιμέρους κομμάτια των προγραμμάτων φυσικά, αλλά που συμβάλλουν στο συνολικό αποτέλεσμα. Μία ερώτηση. Τα ITI θα μπορούσαν ενδεχομένω να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη των στρατηγικών, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών που διαδίδονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση πώς ε, μπορούν ε, τι περαιτέρω κίνδυνοι και επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν αν τέτοια μέσα τα απεφαίνεται να είναι τα καταλληλότερα για ε, κοινωνικό προγραμματισμό στο τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο σε διαφορετικούς τομείς. Οπότε εκεί χρησιμοποιούνται πολλά ταμεία για διάφορες περιφέρειες, διάφορους δήμους. Πώς λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει συγκεκριμένα ένα ITI που αφορά μια μεγάλη περιοχή η οποία ενδεχομένως ε, ανοίξε περισσότερες από μια χώρες. Πιστεύω λοιπόν παρόλα αυτά φυσικά ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν ιδιαίτερα ε, κατάλληλο για τέτοιες στρατηγικές. Ε, εκεί θα πρέπει να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ καλή έκθεση της ε, κυρίας Τόμας, θέλω και εγώ να την ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ε, επενδύσεις ε, σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του κόσμου και των τοπικών φορέων έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν πιστεύω ότι στις περιφέρειες εκείνες ε, ε, αποδίδουν περισσότερα τα μέσα όσο πολλαπλασιάζει το αριθμός τους ή ο αριθμός των φορέων που τα διαχειρίζονται. Το θέμα είναι πώς γίνεται η διαχείριση, όχι πώς είναι αυτοί που την κάνουν. Γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα που διαχειρίζονται αυτά τα εργαλεία. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι τελικοί δικαιούχοι που είναι μικρές μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, τελικά δεν ε, βλέπουν τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα και όταν είναι τόσοι πολλοί μεσάζοντες τελικά χάνεται και η εμπιστοσύνη και επικρατεί μια καχυποψία και μια δυσπιστία. Βέβαια Εντάξει, η ε, δημόσια διοίκηση θέλει ένα περιθώριο ελιγμών ή ένα χρονικό περιθώριο, πράγμα που περιορίζει τη δυνατότητα δράσης των τοπικών ε, οργανώσεων που θα ήθελαν να υποφελούνται από τα μέσα και τα ταμεία αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς γίνεται η διαχείριση στα διάφορα επίπεδα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία το τελικό επίπεδο, ο τελικός δικαιούχος να ξέρει ε, τι γίνεται και να παίρνονται και οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο και να έχουν την περισσότερη επιρροή και το μεγαλύτερο λόγο για το πού θα πάνε τα χρήματα για να πιάσουν τόπο. Τι εννοώ. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φανταστικό, ένα ε, τέλειο μέσο να καλούμε την τοπική κοινωνία να δράσει και μετά να τους ε, υψώνουμε ένα σωρό διοικητικά εμπόδια που να τους αποθαρρύνουμε. Η συγκήτρια επίση. αναφέρθηκε σε κάτι άλλο που θέλω να πω. Υπάρχουν διάφοροι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τοπικές οργανώσεις που δεν μπορούν να εκτελέσουν όλα αυτά τα προγράμματα, να χαράξουν στρατηγική, δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα αντικειμενικά. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα τους διευκολύνουμε και πώς θα τους βοηθάμε σε όλα τα επίπεδα και πάλι. Αν χρειάζεται να γίνει μια διοικητική δουλειά, να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. πολύ. Και τώρα, τελευταίος, ο κύριος Μπούντα βέβαια, εξίσου σημαντικός με τους υπολείπους αλίμων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Δυστυχώ είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο μου. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια και να πω ότι από την περασμένη συνεδρίαση ε, συναντήθηκα με πολλούς εκπροσώπους από τη Ρουμανία και με εκπροσώπους ε, τοπικών ομάδων δράσης και συζητήσαμε αυτά τα μέσα. Και τι ε, μας είπαν αυτοί. Με παρακάλεσαν για το εξή. Χαίρονται που βεβαίως έχουν εργαλεία στη διάθεσή τους, αλλά θέλουν να είναι και λειτουργικά. Η δική μου χώρα έχει γενικά χορτάσει από γραφειοκρατία. Τώρα έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό που ξέρει πώς δουλεύουν οι Βρυξέλλες και ελπίζουμε να τα βγάλει πέρα. Αυτό το θέμα της αποκέντρωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης. για να μπορούν οι τοπικές αρχές να εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας, να τους δίνουμε εμείς τη δυνατότητα. Οι τόποι είναι εκείνοι που ξέρουν τι χρειάζεται ο τόπος τους, δεν θα τους πούμε εμείς. Όταν το σύνολο των φόρων συλλέγονται σε εθνικό, κεντρικό επίπεδο και αν δεν ξαναβλέπουν τα λεφτά αυτά οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων. Γι' αυτό μαστίζει όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στη Ρουμανία. Μπορούν να μας βοηθήσουν λοιπόν όλα αυτά να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Με ιδιωτικές επενδύσεις επίσης, τις οποίες θα προσκαλούμε, θα κινητροδοτούμε και θα ενισχύουμε. Για να τονωθεί η ύπεθρος και η περιφέρεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές τις δυνατότητες για να αναπτύξει ο καθένας την ε, δράση του. Είμαι πεπισμένος ότι τελικά θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε ο καθένας στη χώρα μας για να ε, παρουσιάσουμε αυτά τα εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πριν ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Τόμασιτς, θέλω να ακούσω την απάντηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας απευθύνθηκαν ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Ναι, όντως, ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Συζητάμε για δύο διαφορετικά ε, εργαλεία και τα δύο επιτρέπουν ε, εφαρμογή προγραμμάτων ε, με ολοκληρωμένο τρόπο και υποστήριξη από διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία. Για την τωρινή προγραμματική περίοδο ε, υπάρχουν ήδη κατευθυντηρίες γραμμές, ακόμη και σε στάδιο προγραμματισμού, γιατί ακούσαμε κάτι σχετικό. Για όλα τα στάδια των προγραμμάτων, ακόμη για τον προγραμματισμό, λοιπόν, υπάρχει, υπάρχουν κατευθυντηρίες γραμμές. Για το ο κύριος Φανεστερόη μας ρώτησε συγκεκριμένα ε, σε ποιο ποσοστό ε, θα εφαρμοστούν και ποια θα είναι τα ποσά. 20 ε, κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν το e ε, στα πλαίσια διαφορετικών ε, ολοκληρωμένων στρατηγικών και με διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Τα δύο τρίτα από αυτά τα ε, κονδυλία θα χρησιμοποιηθούν για αστικές στρατηγικές, είναι υποχρεωτικέ εξάλλου στο τωρινό πλαίσιο βάση και των στόχων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή επωνομαζόμενες στρατηγικές άρθρου 7, 16 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ATIs για να υποστηρίξουν αυτές στις ε, ε, στρατηγικές σε αστικές ζώνες τουλάχιστον 5% των επιπρόσθετων πόρων θα διοχετευθούν σε αστικές ζώνες και βλέπουμε ότι προς το παρόν ε, διοχετεύονται για το αστικό περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση και για τις βιομηχανικές στρατηγικές χαμηλής, χαμηλών εκπομπών διοξίδιο άνθρακα. Για το... Υπάρχουν και άλλου τύπου ε, στρατηγικές ε, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. αλλά πάλι σε σχέση με το περιβάλλον και κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου ε, ενδέχεται να αλλάξουν προς ανατολισμό ε, κάποια κράτη-μέλη. Σε σχέση και με τα άλλα τέσσερα ταμεία και συγκεκριμένα για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, τουλάχιστον 17 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές ε, και 1,2 δισεκατομμύρια έχουν ε, στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήδη εκταμιευθεί στα πλαίσια των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης ε, που είναι υποχρεωτικές ε, επιπροσθέτως σε σχέση με το Ταμείο Αλίας γιατί αυτό είναι μια επιπρόσθετη δραστηριότητα και επιπροσθέτως σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι σχετικά νέο στοιχείο ως προς την στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνουμε και φυσικά επειδή είναι μεικτή η διαχείριση των προγραμμάτων με τα κράτη-μέλη θα παρακολουθούμε την εφαρμογή τους, θα δρομολογήσουμε και ε, μελέτες οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες και φυσικά θα συνημερώσουμε για τα πορίσματα για, τα καλύτερα, ε, για τις καλύτερες στρατηγικές, ε, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, για τα Ε, Θα δούμε λοιπόν για τα επιχειρησιακά προγράμματα ποιες στρατηγικές ακολουθούν τα κράτη-μέλη ποιες προτιμούν. Για τις στρατηγικές ε, άρθρου 7 για τις αστικές ζώνες έχουμε και δίκτυο υποστήριξης, γιατί κάποιοι ζήτησαν ε, ε, πρόσθετες κατευθυντήρες γραμμές. Λοιπόν υπάρχει αυτό το δίκτυο και προσπαθούμε τα προβλήματα τις ερωτήσεις σε σχέση με τις αστικές ζώνες, είτε σε σχέση με το ETI, είτε σε σχέση με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ε, να είμαστε σε διαρκή διάλογο και με τα, τις περιοχές και με τις διαχειριστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα ε, μέσα από αυτό το δίκτυο. Ε, το CLLD επίσης ε, συνεργαζόμαστε στενά με άλλα ταμεία, με τα υπόλοιπα τέσσερα ταμεία. Κάνουμε κοινέ εκδηλώσεις, παραδείγματο χάρη το Δεκέμβρη στο Εδιμβούργο. Τέσσερα ταμεία θα συνδιοργανώσουν εκδήλωση όλες οι διαχειριστικές αρχές που έχουν ήδη προγραμματίσει η CLLD θα ε, προσκληθούν, καθώς και τοπικούς φορείς. Κύριος, ε, τώρα ασχολούμαστε με την ε, ενημέρωση και ε, με την ευαισθητοποίηση μέσω των MAs, δηλαδή Managing Authorities, διαχειριστικών αρχών, για ε, το CLD συγκεκριμένα ε, έχουμε και συνεργασία και με την Παγκόσμια Τράπεζα, οπότε διευρύνουμε την προσέγγιση μας και βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο πώς, ε, ποιες γραμμές ακολουθούνται. Με τον ΩΣΑ επίσης συνεργαζόμαστε στενά για τις, το θέμα των αστικών ζωνών και την αλληλεπίδραση υπαίθρου και αστικών κέντρων και υπάρχει μια διαρκής ενημέρωση και διαρκής διάλογος που μας ε, ενδιαφέρει επίσης. Αυτά τα σχόλια έχω να κάνω. Ευχαριστώ. Ε, μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, εισηγήτρια την κυρία Τόμασιτς για να απαντήσει σε ερωτήσεις, να κάνει τελικά σχόλιο, ό,τι θέλει. Ευχαριστούμε. Είπα πως αυτό είναι το πρώτο σχέδιο εκθεσής που υποβάλλω. Ε, έβαλα τα δυνατά μου. Άκουσα από πολλούς και παρατήρησα και εγώ πως χωλένουμε ως προς την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, Ε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές στρατηγικές. Άρα δεν ε, λαμβάνουν όλοι την ίδια ενημέρωση. Χάνουν την εμπιστοσύνη που έχουν λοιπόν στο, στην νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πολλοί ζήτησαν τη σύσταση ενός ε, ε, ανεξάρτητου οργανισμού μιας ε, ενός κεντρικού σημείου επαφής για να ενημερώνονται ή να ε, αναφέρουν ότι υπάρχει κάποια έκνομη δραστηριότητα ή δεν βαίνουν αισίως τα προγράμματα. Δηλαδή, πολλές δυσκολίες μπορούν να αποδοθούν σε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα ήθελα να βελτιώσω την έκθεση και με χαρά θα ε, ενσωματώσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ε, η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου, Τετάρτη, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων για την εδαφική συνεργασία της βέλτιστης πρακτικές και τα καινοτόμα μέτρα. Τώρα... Θα δώσω το λόγο στην υποφαινόμενη, γιατί είμαι εγώ η συγγήτρια να ρωτήσω τους συναδέλφους υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία όταν είναι η πρόεδρος ε, η συγγήτρια κανείς δεν λέει κάτι όχι μου λένε όλοι οπότε περνάω στο ρόλο της συγκήτριας λοιπόν ε, επιτρέψτε μου να μιλήσω στη δική μου γλώσσα στα βουλγάρικα γιατί προτιμώ να μιλήσω τη δική μου γλώσσα Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι ένας από τους τομείς ε, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τα κράτη-μέλη και για το περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η ETS, ε, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ε, διασυνοριακών ε, διεθνών συνεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα θα σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες δικές μου όσον αφορά αυτή την έκθεση. Η παρουσίαση αυτή θα λάβει υπόψη την σπουδαιότητα του ETS ε, και του Interreg. Το ETS ε, αποτελεί ε, σημαντικό κομμάτι της πολιτικής συνοχής και εγώ θα προσπαθήσω να εστιαστώ ε, στην κύρια δομή της εκθεσής μου. Θα σας παρουσιάσω τα κυριότερα θέματα που θα επισημάνω στο κείμενο. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι η προστιθέμενη αξία του ETS και το πώς αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μετά θα περιγράψω τη συμβολή του ΙΤΕΣ για την επίτευξη των στόχων της εδαφικής συνοχής. Τρίτον, το ΙΤΕΣ είναι ένα εργαλείο υποστήριξης της εδαφικής καινοτομίας. Τέταρτον, συμβάλλει στο συντονισμό πολιτικών ε, και στη συνοχή τους Και εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικές οι ευρωπαϊκές ομάδες εδαφικής συνεργασίας. Ελπίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της εκθέσης αυτής θα είναι το θέμα της απλούστευσης του ETC. Ε, αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα για όλους τους τομείς της πολιτικής συνοχής και έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του ETC, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Θα εστιαστώ επίσης ε, στο τι θα γίνει μετά το 2020 και στο πώς θα ενισχύσουμε την δημόσια εμπιστοσύνη και πώς θα προβάλλουμε περισσότερο του ETC, την ETC. Όλα αυτά τα θέματα μπορεί να οδηγήσουν σε ζωηρές συζητήσεις ε, αλλά και να δημιουργήσουν το πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ήτηση. E Ιδιαίτερα στο ρόλο που διαδραματίζει στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε και πολλές άλλες πτυχές Ελπίζω ότι σήμερα σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση θα μπορέσετε και εσείς να μου επισημάνετε επιπλέον ζητήματα. Τώρα όσον αφορά την ήτηση την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και πώς συμβάλλει αυτή στην Στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ήτηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων των περιφερειών, ειδικότερα σε μεθοριακές περιοχές. Η μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχή μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις στο πλαίσιο του ETC, της ETC, καθιστά τις επενδύσεις πιο αποτελεσματικές, πιο στρατηγικά προσανατολισμένες και πιο επικεντρωμένες, ε, κάτι που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Ε, τουλάχιστον το 80% της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ETC καταχωρείται σε τέσσερις ε, τομείς κλειδί καινοτομία και έρευνα, ψηφιακό θεματολόγιο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δεν είναι τυχαίο. Ε, ο νέος σχεδιασμός ε, της, των προγραμμάτων βάση επιδόσεων θα βοηθήσει να χρηματοδοτηθούν περισσότερα προγράμματα μέσω της η οποία αναζωογονείται ως ένα νέο μέσο ε, της πολιτικής συνοχής μέσο το οποίο θα συμβάλλει ε, σε καλύτερα αποτελέσματα, σε πιο αποτελεσματικά μέτρα ε, που θα βοηθήσει για μεγαλύτερη συνοχή. Στην έκθεση μου επίσης θέλω να επισημάνω την υποστήριξη και συμβολή της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας υπό την οποία η ETC μετατράπηκε ξανά σε προτεραιότητα η Προεδρία συνέδεξε πολλά έγγραφα για το θέμα αυτό, τα οποία παρουσιάστηκαν ε, σε πολλές και διάφορες ε, ειδικά αφιερωμένες συναντήσεις. Έτσι λοιπόν η Λουξεμβουργιανή Προεδρία άνοιξε το δρόμο για ένα όραμα για την περίοδο μετά το 2020 βάσει μιας ανάλυσης επιδόσεων ε, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου καθώς και σε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των αλλαγών της ΣΥΤΙΣΗ εντο εντός περίοδου 2014-2020. Επ' αυτού η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μια εκτίμηση αντικτύπου το 2016 μάλιστα και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, επίσης πρόκειται να εκδώσει μια γνωμοδότηση για τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δική μου έκθεση θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για να εστιαστούμε περισσότερο στις επιδόσεις, να επικεντρωθούμε στις επιδόσεις ε, και στο να ενισχύσουμε τον προπολογισμό για την εδαφική συνεργασία. Η χρηματοδότηση τη εδαφική συνεργασία πρέπει να προσαρμόζεται καλύτερα σε διάφορε περιφέρειες, σε διάφορε περιοχέ. Η πιο καλά προσαρμοσμένη χρηματοδότηση είναι κάτι που ήδη συζητείται εντό τη ε, Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη εδώ. Ε, αλλά μπορούμε να εμβαθύνουμε και περισσότερο όσον αφορά, για, να δούμε τι θα κάνουμε στην περίοδο μετά το 2020. Πρέπει να δούμε πώς θα ε, εξολογήσουμε τον προπολογισμό και πώς θα μπορούμε να δίνουμε περισσότερα κονδύλια στα μέσα που ε, στοχεύουν στην εδαφική ε, συνοχή. Είναι σημαντική και η συλλογή και η ανταλλαγή ε, στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών τόσο τα κράτη-μέλη όσο και οι περιφέρειες όσο και ε, οι θεσμοί θα πρέπει να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω μέσων όπως το Interact και το ESPON ή να αξιοποιούν δεδομένα που παρέχει η Eurostat. Όσον αφορά τη συμβολή της ε, ETC στην επίτευξη των στόχων της εδαφικής συνοχής, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εδαφικό θεματολόγιο και την πολυκεντρική προσέγγιση για τη δημιουργία νέων εδαφικών μονάδων πέραν των εθνικών συνόρων. Μέτρα τέτοιου τύπου πρέπει να υιοθετηθούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ε, πολιτών που μένουν σε μεθοριακές περιοχές. Ε, έχουν αναλυθεί διάφορα σενάρια και υπάρχει ένα όρομα για την περίοδο μετά το 2020 και βάσει αυτών των πληροφοριών εμείς θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ε, ότι η εδαφική συνοχή και η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να βασιστούν σε μια πολυκεντρική προσέγγιση των ευρωπαϊκών εδαφών. Η ΤΣΥ επίσης είναι σημαντική όσον αφορά τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Ο δεσμό είναι ισχυρό μεταξύ τη εδαφική συνεργασία και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η εδαφική συνεργασία ε, προφανώ ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Τέλο, και εξίσου σημαντικό, πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη περισσότερης συμπληρωματικότητα και βελτιωμένη συνοχή μεταξύ κεντρική εδαφική συνεργασία και του εθνικού επίπεδου. Η εθνική συνεργασία, η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να ε, συμπεριληφθεί και σε άλλα προγράμματα και μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό στοιχείο της εκθεσής μου θα είναι ο ρόλος της ETC, η στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας. Ειδικότερα υπό τα προγράμματα Interreg προσδιορίζονται οι τομείς ε, όπου οι περιφέρειες, οι χώρες ε, ε, και διάφοροι εταίροι θα πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική η επίτευξη της έξυπνης εξειδίκευσης η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα μπορούσε να, χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ως εργαστήριο ε, επόσης ε, καινοτόμων ε, προγραμμάτων σε πολλούς τομείς θα μπορούσαν αυτά μάλιστα να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα μέσα και σε άλλα προγράμματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία διασυνοριακών ερευνητικών εγκαταστάσεων διασυνοριακών ερευνητικών προγραμμάτων και διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τη διαχείριση και το συντανισμό, αλλά και όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Εδαφικής ε, Συνεργασίας, ε, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ε, διοίκησης και συντονισμού. Θα πρέπει να επιδιώκεται συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα ενδεχομένως και συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Κομισιόν θα πρέπει να προβεί σε κάποια αξιολόγηση της συνοχής και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της, ε, των προηγούμενων προγραμματικών περίοδων. Επίσης θα πρέπει να δώσει κάποια ε, πρόβλεψη ε, εκτιμήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η απλούστευση είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την εδευτική συνεργασία. Η απλούστευση είναι κάτι αναγκαίο. Τόσο στους τομείς ε, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ε, του κανονισμού κοινών διατάξεων αλλά και όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές. Πρέπει να παρέχεται με περισσότερη τεχνική υποστηρίξη και πρέπει να εφαρμοστεί και ηλεκτρονική διαχείριση στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά πιο ευρέως και επίσης πρέπει να χρησιμοποιούμε και μέσα όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις και εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και πάλι στον τομέα της ε, εδαφικής συνεργασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι στο τελευταίο, στην τελευταία συνέντευξη του Συμβουλίου η Λεξομβοριανή Προεδρία πρότεινε την εφαρμογή ενός νέου ειδικού μέσου επίλυσης διαφορών μεταξύ εταίρων, μεταξύ κρατών μελών για θέματα εδαφικής συνεργασίας ειδικότερα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομάδων εδαφικής συνεργασίας. Όλες αυτές ε, οι δυνατότητες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω εφόσον συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, αφού μιλάμε για ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, πέραν της ε, τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, θα πρέπει να ενισχύσουμε, πιστεύω, το ρόλο της Interreg να προβλέψουμε καλύτερο συνδανισμό, περισσότερη καινοτομία, προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και ανάπτυξη στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης ε, τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και μεταξύ ε, περιφερειών. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα επίσης το οποίο θα ήθελα να επισημάνω στην εκθεσή μου τη σπουδαιότητα και την προβολή της εδαφικής συνεργασίας. θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις ε, στα προγράμματα ειδευτικής συνεργασίας. Αυτές είναι οι πρώτες ε, ιδέες ε, που έχω να σας παρουσιάσω όσον αφορά την έκθεση αυτή για την ειδευτική συνεργασία. Και περιμένω τα σχόλιά σας και να ζητήσω από τον κύριο συγητή, τον κύριο Χίτμαν, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του εγγράφου. Ελπίζω να το λάβουμε συντόμως. η εδαφική συνεργασία είναι κάτι που ενδιαφέρει τους δικαιούχους ε, τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα ε, εργαλείου που ε, λατρεύουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η κοινωνικοί εταίροι, και πολλά προγράμματα εφαρμόζονται πραγματικά στη βάση, υλοποιούνται για να ρυθμίσουν πολύ πρακτικά προβλήματα. που ε, καμιά φορά ε, φαίνεται να μην είναι τόσο σημαντικά όταν κάποιος θα εξετάζει από πλευράς ε, από τις Βρυξέλλες το ETS, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, είναι στοιχείο κλειδί της ε, πολιτικής συνοχής ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που θέλετε, Πρόεδρε, να ε, δώσετε έμφαση στην διάδοση των αποτελεσμάτων τέτοιων προγραμμάτων, διότι παραγνωρίζεται ε, η σημασία του συχνά, παρότι έχουν μεγάλο ειδικό βάρος για τις ε, κοινότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε μεγάλη ευελιξία σε σχέση με την χρήση αυτού του εργαλείου. Νωρίτερα ε, είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε περιβαλλοντικά προγράμματα, στον τουρισμό, στις υποδομές, ε, στις ανταλλαγές ε, των, για τους νέους. Είναι ε, εκπληκτικό αυτό το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και θα πρέπει να διαδίδονται τα αποτελέσματά του διότι είναι εξαιρετικά επιτυχημένο. Οι βέλτιστες πρακτικές λοιπόν θα πρέπει να διαδίδονται ούτως ώστε να υποφελούνται και οι μελλοντικοί δικαιούχοι. Ένα πρόγραμμα παραδείγματο χάρη που εφαρμόζεται από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν όλες να υποφεληθούν από ε, παρελθούς πρακτικές και ε, χαίρομαι επίσης που αναφέρατε, προαναγγείλατε απλούστευση του συστήματος. Στην Πολωνία έχω προσωπική εμπειρία για την περιφερειακή συνεργασία και αυτοί που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων αξίζουν το σεβασμό μας, διότι κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό, πρέπει να προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο και Είναι πολύ καλό να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εμπειρίες που έχουμε για την υλοποίηση των μελλοντικών προγραμμάτων. Αυτοί που ε, είναι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμβάλλουν ναι, και στην ε, κατάρτιση των προγραμμάτων Αναφερθήκατε επίσης, ε, Πρόεδρε, στο ότι το Interreg θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιτέλους ως εργαλείο της εδαφικής συνεργασίας. Έχει παγώσει προς το παρόν αυτή η ιδέα και δεν εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Ίσως όχι διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, αλλά διότι απουσιάζουν οι συστημικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων που ζητούν ε, οτά σε διασυνοριακό επίπεδο. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε δε και μια πρωτοποριακή προσέγγιση σε σχέση με το, την εδαφική συνεργασία. Δηλαδή, πέρα από τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, να κάνουμε ένα επιπρόσθετο βήμα και να δούμε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το στοιχείο της έρευνας και ανάπτυξης μέσα στην έκθεση για να προχωρήσουμε περισσότερο. Ίσως στο μέλλον θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε ε, κάποιες επιχειρηματικές λύσεις που έχουν μια διασυνοριακή διάσταση. Η συνεργασία αυτή υπάρχει, όμως ε, ενδεχομένω δεν λαμβάνουν αυτές, αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια άμεση επιδότηση. Κυρίως τώρα που πλήττονται πολλά από υψηλά ποσοστά ανεργίας, θα έπρεπε ίσως να ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις, παραδείγματος χαρή, μεθοριακών περιοχών, τα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα θα μπορούσαν να ε, συλλειτουργήσουν με επιχειρηματικά σχέδια που ε, δημιουργούν θέσεις εργασίας και χάρη στα οποία αποφεύγουμε ε, την μαζική μετανάστευση των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ελπίζω λοιπόν να είναι πλούσια η συζήτηση που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και Πρόεδρε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης η έκθεσή σας. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Κυρία Μπρέσου θέλει το λόγο. Θα ήθελα μόνο να πω πως η κυρία Νταντσίλα δυστυχώς απουσιάζει και Μου έστειλε γραπτό στη θέση της σκιώδης εισηγήτρια. Ε, Έχουμε σε διαδικασίες όπως βλέπετε, αλλά είναι επειδή που είναι συνεδρία στη Δευτέρα και δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος ε, Βανίτεμπορκ, ο κύριος Βαν Μίλτεμπορκ θα πάρει το λόγο. Ε, ναι, να τον πάρω, αφού μου το δίνετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρότασή σας για τη μέθοδο εργασίας με την έκθεσή σας είναι πολύτιμη. Έχω δύο σημεία. Uh, το πρώτο είναι η διασυνοριακή ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να λυθεί και να το εξετάσει και η έκθεσή μας, γιατί πιστεύω ότι πολλοί Ευρωπαίοι είναι ταλαντούχοι, είναι πρικισμένοι, αλλά δεν μπορούν να ε, ασκήσουν ε, αυτές τις δεξιότητες τους από την άλλη μεριά των συνόρων γιατί υπάρχουν βαριές διαδικασίες, προβλήματα εθνικού ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε ε, την κινητικότητα των εργαζομένων. Ξέρω ότι θα έρθει το πακέτο με μέτρων της Επιτρόπου Τέισεν, αλλά έχει και μεγάλη σχέση με την εδαφική συνεργασία. Το δεύτερο έχει να κάνει με την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου και τη διαχείριση των προγραμμάτων τους κανόνες. Εγώ συζητώ ε, με επιχειρηματίες για το Ιντερεκ και το πρώτο που μου λένε είναι ωραίο είναι αν θες να πάρεις μια πιστοποίηση ε, ως ειδικό της διοίκησης για το πώς θα χειρίζεσαι λογαριασμού, θα εκαθαρίζει λογαριασμού για το πώ θα λύγει τον κόσμο σε μια κόλλα χαρτί. Αν θε να συζητά με πολλού ελεγκτέ και οικονομικού ελεγκτέ για τη διαχείριση, αν δεν είναι όμω αυτή η βασική σου δουλειά, αν δεν είσαι λογιστή αλλά επιχειρηματία και θε να στήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια νεοφυή, και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσεις πλούτο, ανάπτυξη και δουλειέ ε, καμιά φορά φρακάρες σε όλη αυτή τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπου απαιτούνται και άλλα προσόντα από τον να είσαι καλός επιχειρηματίας. Πρέπει να είσαι αρκωτός λογιστής περίπου. Πώς μπορούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων, ιδιαίτερα όταν έχουμε την Ευδαφική Συνεργασία και το Ιντερεκ και τη χειριστική αρχή μπορεί να είναι σε άλλη χώρα. Α πούμε στι κάτω χώρε όταν μιλούμε για ένα πρόγραμμα Interreg, θα πρέπει να πάμε στη Λίλη, Νορ Πάντε Καλέ, στη Γαλλία. Και φανταστείτε τι θα γίνει μετά τι γαλλικέ περιφερειακές εκλογές. Αν κερδίσει εκεί το εθνικό μέτωπο και διαχειρίζεται τα περιφερειακά ταμεία, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Βέβαια, δεν ήθελα να πω αυτό εγώ, εμπαρόδο το λέω. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα απλουστεύσουμε τις διαδικασίες για τη διασυνεργική συνεργασία. Βεβαίως μπορούμε να την εθαρρύνουμε, αλλά να είναι πιο απλοί οι κανόνες για να δουλεύει το σύστημα και να μειώσουμε το γραφειοκρατικό, το διοικητικό κόστος. Γιατί οι επιχειρηματίες, οι πανεπιστημιακοί δεν ε, επιλέγουν να υποβάλουν ε, αίτηση για να τους νίξουμε στο χάρτο βασίλειο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάνα. Στα αγγλικά. Θέλω και πάλι να ζητήσω συγγνώμη ε, από το εξ του του Σιγητού που κολλείται και μου έχει στείλει τις απόψεις του. Καλώς όρισε πάρα πολύ και χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, όχι μόνο ε, επειδή κλείνει 25 χρόνια το Ιντερεκ, το Συμβούλιο ενέκρινε κάποια συμπεράσματα, το ακούσαμε ήδη πριν από 10 μέρες. Η Ευρωπαϊκή ε, η εδαφική συνεργασία είναι ένα μόνο εργαλείο και μέσο στην ε, πολιτική συνοχή. συνοχής. Όσο περισσότερο διαρκεί μια διασυνοριακή συνεργασία, τόσο πιο έντονη γίνεται και τόσο πιο λίγο χωρίζει το σύνορο της δύο χώρες. Γι' αυτό έχει σημασία να δίνονται επαρκείς και αποτελεσματικοί πόροι στην Ευρωπαϊκή ε, Εδαφική Συνεργασία στο σημερινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, δεν ισχύει αυτό. Το Συμβούλιο μείωσε την αντίστοιχη ε, θέση του προπολογισμού, ενώ το Κοινοβούλιο ήθελε να την αυξήσει. Υπάρχουν προγράμματα όπως είναι θεματική συγκέντρωση και η προσήλωση ε, και ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Η εδαφική συνεργασία παίζει σημαντικό ρόλο επιπλέον στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν κονδύλια να πάνε και εκεί. Ο κύριος Μπόνις Χόπε, ο ε, σκιώδης μας, ε, με χαρά να συνεργαστεί. Έχει τεράστια εμπειρία, πρέπει να ξέρετε, στην εδαφική συνεργασία, διότι 20 χρόνια ήταν δήμαρχος μιας παραμεθόριας πόλης και θέλει να επικεντρωθεί σε τρία ζητήματα. Πρώτον, πρακτικός αντίκτυπος της εδαφικής συνεργασίας στην πραγματική ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών. Το δεύτερο είναι ορισμός της εξαιρετικής ιδιαίτερης ποιότητας αυτής της συνεργασίας που διαφέρει από τα κλασικά προγράμματα της συνοχής και το τρίτο που θέλει να τονίσει είναι ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής στο σύνολο. Pardon, in uh, particular. Thank you. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Thank you very... Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε Αντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εδαφική συνεργασία ε, είναι ένας από τους στόχους των διαρθρωτικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων Μιλάμε για μεγάλε ε, δαπάνες, πολύ σημαντικές αυτή την ιστορική στιγμή, ώστε να ενθαρρύνουμε τι ε, εδαφικές περιοχές διαφόρων κρατών μελών να συνεργαστούν με ανταλλαγή εμπειριών. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική συνοχή, πολιτική συνοχής, ε, ώστε να επιτευχθούν ε, οι στόχοι. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποιες περιοχές ε, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και στη συνεργασία μεταξύ περιφερειών θα μπορούσε να είναι πολύτιμη. Η εδαφική συνεργασία και η, κυρίως η παραμεθορία συνεργασία είναι σημαντική, οπότε πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιοχής, μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να διαφυλάσσονται, όπως και σε άλλες ε, περιπτώσεις. Δεν πρέπει να καταλήγουμε ποτέ την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Εγώ είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία με ως εισηγήτρια και με τους σκιώδεις εισηγητές ε, θα είναι ιδιαίτερα συνεργατική και επικοδομητική. Εγώ είμαι αναπληρώτρια σε αυτή την επιτροπή και ελάχιστες φορές έχω παρέμβει, αλλά είμαι βέβαιη ότι αυτό θα αποτελέσει μια ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα τους συναδέλφους και να ξεκινήσουμε μια πραγματικά πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βανίσταλ Ροέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνεχίζοντα από εκεί σταμάτησε ο προλαλή σα ε, του ΕΛΚ Χέτμαν, θέλω να πω το εξή. Στην παρουσίασή σας τονίσατε πάρα πολύ και ρίξατε το βάρος στις μελλοντικέ προοπτικές. Στο μέλλον γενικότερα, όχι μόνο βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα. Το μέλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά. Γιατί απογοητευτήκαμε τόσο πολύ στην, ε, συζήτηση, στην, στην, στην, έκτη έκθεση για τη συνοχή. Η εδαφική συνεργασία, η εδαφική συνοχή είχε γίνει υπολεπτομέρεια. Και το Κοινοβούλιο καλά θα κάνει και καλά κάνει που του δίνει νόημα και περιεχόμενο στραμμένο προς το μέλλον. Να μην κοιτάμε μόνο τι γίνεται στην πράξη, αλλά τι γίνεται και προοπτικά. Ε, είναι τεράστιο αυτό το βήμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν κοιτούμε, ε, κοιτάξουμε πώς έχει η σημερινή κατάσταση, τώρα ξεκινάει η περίοδος 2014-2020. Είχαμε ε, δύο καλά χρόνια να μην πω δύο χαμένα χρόνια, ε, προσπαθούμε να στήσουμε από την αρχή τους κανονισμούς με τα συμβόλαια εταιρική συνεργασίας και τα επιχειρησιακά και μόνο ε, από τη μετάφραση. Ε, οπότε δεν θα έχουμε πια χρόνο για να δούμε τι θα γίνει μετά το 2020. Αν θέλουμε αλλαγέ, αυτό θα πρέπει να γίνει το 2018 και μάλιστα στα μέση του 2018 να έχει ολοκληρωθεί για να υπάρχει μια ε, νέα πρόταση και χαίρομαι πάρα πολύ. Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό που πρωτοστατεί το Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Το Κοινοβούλιο ήταν δυσαρεστημένο. Θυμάστε την έκθεση Deutsch για τη συνοχή, για το τι γίνεται με την εδαφική συνεργασία. Αυτό είναι και παραμένει ε, ουσιαστικότατο. Και να δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο. Μας είπατε ότι πήγατε ίδια στο Λουξεμβούργο. Η εδαφική διάσταση είναι κάτι που δεν αφισβητεί κανένα κράτος μέλος. Είδαμε τι έγινε πριν από 15 μέρες και στην Επιτροπή Περιφερειών που συνεδρίασε από κοινού ε, με εκπροσώπους των παραμεθόριων περιφερειών και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη απειλή. Κοιτάξτε τι γίνεται με το Σέγγεν, υφίσταται πίεση. Μα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων παρακαλώ λένε να ζήσουμε τώρα με ένα μίνι Σέγγεν. Κάπως να το συρρυκνώσουμε. Όχι, θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ε, ότι ποτέ πια τέτοια πράγματα το βλέπουμε ήδη στα σύνορα. Η εδαφική συνεργασία από εκεί κρίνεται ε, και ε, από εκεί θα δοκιμαστεί και θα αποτύχει, θα επιτύχει. Εμείς θέλουμε να ρίχνουμε σύνορα, να σβήνουμε σύνορα, όχι να σχεδιάζουμε και να ζωγραφίζουμε και άλλα στους χάρτες. Κοιτάξτε πώς έχει η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη και η εδαφική πολιτική και η περιφερειακή πολιτική είναι κομβική και κεντρική σημασία. Πολύ καλό αυτό το μήνυμα λοιπόν που στέλνουμε και προσβλέπω και στη συζήτηση. Ό,τι και να γίνει σε άλλους τομείς πολιτικής, ε, χρειάζεται πολιτική συζήτηση για την εδαφική συνεργασία και τη διασυνοριακή, η οποία κερδίζει νομίζω σε σημασία. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και με χαρά περιμένω να δω και κανένα κειμενάκι. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμένα θα με ενδιαφέρε ιδιαίτερα να δω πώς θα ασχοληθείτε με τις πτυχές της καινοτομίας στον τομέα αυτών. Όπως μας υπενθυμίσετε μάλιστα κι εσείς, ε, ξαφνικά σκεφτόμαστε ξανά αυτό το μέσο μετά από 25 χρόνια χρήσης. Είναι πολλά τα ε, 25 χρόνια. Εγώ ανέκαθεν ζούσα σε παραμεθόρια περιοχή και ανέκαθεν υποστήριζα τις πολιτικές ε, εδαφικής συνεργασίας και διασύνορικες συνεργασίας. Αλλά όπως γνωρίζετε, η εδαφική συνοχή ε, διαιρείται σε τρία μέσα. Ένα που αφορά τις παραμεθόριες περιοχές, ένα άλλο που αφορά τις περιφέρειες και ένα άλλο το οποίο δημιουργεί δίκτυα ε, μεγαλύτερων αποστάσεων μεταξύ περιφερειών, εικονικά θα έλεγα δίκτυα που δεν λαμβάνουν υπόψη, δεν εξαρτώνται από τις ε, πραγματικές ε, αποστάσεις, φυσικές αποστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε το ποιο ήταν το προϊόν αυτών των μέσων όσον αφορά την πραγματική συνοχή ειδικότερα στις παραμεθορίες περιοχές γιατί ξέρετε ίσως να έχει επιτύχει περισσότερα το Σέγγεν το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια έντονη κρίση λόγω των, της δραματικής επικαιρότητας αλλά πραγματικά ίσως το Σέγγεν να έκανε περισσότερα για να εκμηδενήσει τις αποστάσεις από ότι τα μέτρητα μικροπρογράμματα που περισσότερο μεθοδολογικά ήταν παρά επικεντρωμένα στην τοπική ανάπτυξη. Τώρα λοιπόν για να εξελιχθεί το μέσο αυτό θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε ένα μέσο το οποίο θα αναπτύσσει περισσότερο πολιτικές παρά μεθόδους. Το σημαντικότερο μάλιστα θα είναι να δούμε πόσες ευρωπαϊκές ομάδες συνεργασίας έχουν δημιουργηθεί βάσει του προγραμματισμού που γίνεται δύναμη αυτών των μέσων. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο αυτά τα μέσα είναι ακόμα ωφέλιμα. Αν υπάρχει ήδη μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Χρειάζεται να υπάρχουν τέτοια μέσα ενδιάμεσα όταν υπάρχει μακροπεριφερειακή στρατηγική. Δεν θα ήταν καλύτερο τέτοιοι πόροι να μετατοπιστούν σε μεγαλύτερης διάστασης προγράμματα. Το θέμα λοιπόν του πώ θα εφαρμόσουμε καινοτομίε, δεδομένου ότι μεταξύ παραμεθορίων περιοχών ε, έχουν συζητηθεί πολλά, αλλά όχι παντού. Σε ορισμένα μέρη, ναι βέβαια, αλίμονο. Σε ορισμένα μέρη τέτοια προγράμματα πραγματικά οδήγησαν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ε, δήμων, ε, παρεπιστημίων, δημιούργησαν κοινά κέντρα ερευνών, κοινά νοσοκομεία κτλ αλλά πρέπει να δούμε πού ε, υπήρξαν τέτοια αποτελέσματα και πού όχι. Δηλαδή που υπήρξε χρηματοδότηση πολλών μικρών έργων χωρίς τελικά να είδαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την ε, εδαφική ανάπτυξη και την χρήση των ε, βασικών κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Έχουμε το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο συνοχή. Χρησιμοποιούνται όντω από κοινού αυτά τα ταμεία στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Γιατί αν όχι, ε, ε, δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες ε, Πρέπει να δούμε δηλαδή και τι μαθαίνουμε, τι δίδαγμα αποκομίζουμε μετά από τη χρήση αυτών των πόρων. Ε, αυτά που ουσιαστικά χρηματοδοτούν τη δημιουργία δικτύων μεταξύ διαφόρων ε, σημείων της ε, Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Τι αποτελέσματα συγκεκριμένα έδωσαν Ουσιαστικά πρόκειται για μέσα που χρησιμοποιούνται για να βρει κανείς ε, συνεργάτες ε, ε, για κοινά προγράμματα ή μήπως το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να προγραμματίσουμε το μέλλον θα ήθελα να βασιστούμε σε μια ανάλυση των πραγματικών αποτελεσμάτων στον τομέα αυτών πέραν των ε, καθυσχαστικών σχολείων διότι αν τελικά ανακαλύψουμε ότι είναι ελάχιστη συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές ε, αυτό θα δημιουργήσει κάποιες αμφιβολίες για τη χρησιμότητα τελικά αυτών των ταμείων ε, στο παρελθόν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν πώς να το πω, να μην τα θεωρούμε τα πρώτα δεδομένα. Πρέπει να κάνουμε και καμιά ερώτηση που και που λίγο πιο στοχευμένη, ε, λίγο πιο δύσκολη. Πραγματικά να ψάχνει να βρει τι γίνεται στο βάθος ε, ε, σε μια Ευρώπη που είναι εξοπλισμένη με τόσα μέσα κατάργησης των συνόρων τα οποία όμως επανεμφανίζονται ξαφνικά μόλις ε, κάποιος εξωτερικός παράγοντας ε, ε, οδηγήσει σε εθνικιστικές αντιδράσεις. Έχω λοιπόν κάποιες ανησυχίες και θα ήθελα να συμπεριλάβετε και κάποια αμφιβολία σε αυτή την έκθεση κυρία Πρόεδρε πέραν φυσικά της σωστής σκέψης φυσικά ότι είναι, υπήρξε κάποια χρησιμότητα υπήρξαν χρήσιμα αυτά τα μέσα στο παρελθόν είναι ακόμα με ποιο τρόπο. μήπω πρέπει να τα επανασχεδιάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που αργοπόρησα. Ήμουν στη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας και δυστυχώς δεν άκουσα την παρουσίασή σας. Διάβασα όμως τα έγγραφα. Ακούσαμε ε, τα περί απλούστευσης ε, της διοίκησης και της ανταλλαγής ε, των βελτίστων πρακτικών για την εδαφική συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό να ρωτήσω. Έχουμε κάποιους μετρήσιμους στόχους Με την εφαρμογή του ειδικού κανονισμού, για πρώτη φορά βασίζεται η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία σε συγκεκριμένους κανόνες. Το επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται στην ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, όπως είπε η κυρία Μπρέσου. Ε, επίσης θα ήθελα να επικροτήσω το στόχο ε, για που έχουμε για τις καινοτόμες λύσεις και νομίζω ότι θα μπορούσατε να το συνδυάσετε και με το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα που θα προτείνετε. Ευχαριστούμε κύριο Σπουδά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με συντομία να σας πω το εξής η εδαφική συνεργασία και συνοχή είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να συζητούμε για Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχει εδαφική ε, συνεργασία. Το είπε και ο κύριος Βανίστεροι. Θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Πού θέλουμε να φτάσουμε, ποιος είναι ο προορισμός μας. Να καταλάβουμε από πού κινούμε σήμερα τι δεν λειτουργεί σήμερα σωστά, τι δεν πάει καλά. Το είπε και ο κύριος Πόλτσακ. Οι στόχοι μας, ορισμένοι τουλάχιστον, πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ε, ότι θέλουν ε, να απλουστευτούν ε, οι διαδικασίες και η πρόσβαση. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Εγώ ε, το πρωί συνάντησα γιατρούς, πανεπιστημιακούς και μου είπαν πόσο δύσκολο είναι να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουν τέσσερις ε, προγράμματα στη ΣΥΠΑ, τρία στην Ινδία, δύο στην Κίνα. Αλλά στην Ευρώπη κανένα. Για ποιο λόγο. Και αυτό ισχύει και για την Επιτροπή Γεωργίας και για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τα δικά μας θέματα. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα κονδύλια. Γιατί είναι τόσο βαριές και δύσκολες οι διαδικασίες. Ποιες λύσεις μπορούμε να βρούμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και να καταλήξουμε στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψε. Um, yes. Ευχαριστώ. Ναι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το υλικό που πρόκειται να λάβετε. Το 2016 θα έχετε την ε, post, ε, ex post αξιολόγηση για την περίοδο μέχρι το 2013. Δηλαδή θα έχετε υλικό για να τροφοδοτήσετε τον προβληματισμό σας για το μέλλον και για την ε, επερχόμενη περίοδο. Το η περίφημη έκθεση του άρθρου 16 που είναι, ε, προβλέπεται στον κανονισμό για τις ειδικέ διατάξεις ε, σύντομα θα δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχετε ε, μια καλή εικόνα για τον προγραμματισμό του προγραμμάτων την για την περίοδο 14 20 για πρώτη φορά στην ιστορία όπως είπε και η Πρόεδρος δεν έχουμε διασυνοριακά, διαπεριφερειακά δεδομένα. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε τη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου για το πώς ε, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διάσταση του ζητήματος, όχι μόνο για τα πρόγραμματα Interreg, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι περιοχές ε, την ένταση, ε, την, το, το, το εύρος της συνεργασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε αν ήταν χρήσιμα και αποτελεσματικά ή όχι τα προγράμματα Interreg ή αν δεν, ε, τελικά δεν ε, υπάρχει μια χρηστή διαχείριση των ε, κονδυλίων σε διασυνοριακό επίπεδο. Μέχρι στιγμή δεν είχαμε τέτοια δεδομένα στη διάθεσή μας. Στις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε και μια διασυνοριακή επισκόπηση της κατάστασης μετά από πρωτοβουλία της Κορίνα Κρέτσου. Ο πρώτος πυλώνας είναι να γίνει απολογισμός των ε, εμποδίων που ε, εξακολουθούν να, ε, εμποδι... να στα οποία εξακολουθούν να προσκρίνουν η περιφερειακή, διαπεριφερειακή συνεργασία ε, και μετά την διάμεση έκθεση το 2011 προέκυψε με σαφήνεια ότι όποια και αν είναι τα κονδύλια που έχουμε, όποια και αν είναι η πρικοδότηση του ίντερνετ και δεν τοποθετούμαστε εδώ αν πρέπει να αυξηθεί, να μειωθεί σε σχέση με σήμερα, όποια και αν είναι αυτή η πρικοδότηση, θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες ε, ως προς ε, και τα ελαττώματα αλλά και το δυναμικό κάθε, ε, κάθε τομέα ε, προγραμματισμού. Ε, το Φεβρουάριο του 2015 ασχολήθηκε με αυτό το θέμα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε μια ισχυρή βάση που να βασίζεται σε στοιχεία και τεκμήρια για τη μελλοντική μας αξιολόγηση. Ε, από εκεί ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και ήθελα να προσθέσω αυτά τα στοιχεία στη συζήτησή σας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε ε, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Ευχαριστούμε ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρατηρήσεις της. Μπορώ να σας πω πως Ε, λόγω της κατάστασης γίνεται λόγω και πιο ενδιαφέρουσα η έκθεση επίσης. Όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδουν ε, αυξανόμενη σημασία στην ε, εδαφική συνοχή και συνεργασία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και ε, προσβλέπουμε την στην επόμενη σύσκεψη με τους σκιώδεις εισηγητές. Σβήνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου, δυστυχώς. Δεν ακούγεται. Επανέρχεται. Τώρα θα ε, ασχοληθούμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την εφαρμογή των θεματικών στόχων για την επίρρωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Η κυρία Νταμάτο είναι η συγγήτριά μας. Έχουμε κάποιους από τους κοιόδης παρόντες, άλλους πάλι όχι. Ε, αλλά είναι ε, ρηξικέλευτη η σημερινή συνεδρία από ό,τι βλέπουμε για την παρουσίαση δηλαδή, των θέσεων των σκιωδών εισηγητών. Είχαν πολλές καινοτομίες. Θα ήθελα να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το αντικείμενο της έκθεσης είναι η εφαρμογή των, ε, του στόχου 3 στα συγκεκριμένα προγράμματα και ε, επίσης οι, ε, οι εφαρμοστικοί κανόνες, τους εφαρμοστικούς κανόνες πρόκειται για έκθεση υλοποίησης. Είναι η πρώτη ε, για το 2015. Η κυρία Νταμάτο για, τα, για την αρχική παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπω γνωρίζετε, όπως μόλις, είπε η Πρόεδρος, αυτή είναι η πρώτη έκθεση υλοποίησης εφαρμογής της Επιτροπής μας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ζητείται τέτοια έκθεση λόγω του ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων ήδη σε αυτή την αρχική φάση. Είναι θεμελιώδη σημασία να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο τα προγράμματα αυτά αποτυπώνουν το πνεύμα συμφωνίας και συνεργασίας και τις αρχές του κανονισμού. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια υπήρξε η θέση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά πόσο υπήρξε ή όχι πραγματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις προκριματικές φάσεις. Προκριματικές φάσεις. Αλλιώς υπάρχει κινδύνος τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά σε προχωρημένα στάδια του προγραμματισμού που θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα και λόγω των οποίων θα ένταθει η δυσπιστία ε, ενώπιον των θεσμών που εμείς εκπροσωπούμε. Η επιλογή ε, Καταρχά οργάνωση του θεματικού στόχου της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οφείλεται στο ρόλο τους στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ξέρουμε ότι το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες Ξέρουμε επίσης ότι ο εξυγχρονισμός της οικονομίας, ειδικότερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή της προγραμματικής περίοδου, αλλά ήδη μπορούμε να εξάγουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, χάρη στην παρακολούθηση από την Κομισιόν. Ε, αυτή η παρακολούθηση των συμφωνιών εταιρική σχέση και των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά του πόρου που έχουν κορυφθεί και την ποιότητα του προγραμματισμού. Κατά πρώτο λόγο, ο στόχος 3 δεν προέβλεπε συστηματική χρήση μιας στρατηγικής εφιούς εξειδίκευσης. Καλό θα ήταν λοιπόν να επαληθεύσουμε κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του προγραμματισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να επενδύουν λιγότερα σε κοινοτόμες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζουμε, οι ευφυής ανάπτυξη απευθύνεται σε πολλούς ε, τομείς και στους παραδοσιακούς αντιθέτως. Οπότε θεωρούμε ότι το Joint Research Center της ε, Σιβήλης ε, εφαρμόζει κάποιες πλατφόρμες θεματικές. Θέλω να δούμε κατά πόσο τα μέσα της χρηματοοικονομικής τεχνικής έχουν εισαχθεί στον προγραμματισμό, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκαν παντού αποτελεσματικά στην προηγούμενη πραγματική περίοδο και δεν θέλουμε να συμβεί το ίδιο και σε αυτή τη νέα περίοδο. Επίσης ε, διερωτόμαστε κατά πόσο η απλούστευση, μια από τις βασικές αρχές της νέας προγραμματικής περίοδου εφαρμόζεται πραγματικά στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά απαντούν δυσκολίες ε, πρόσβαση στα κονδύλια τόσο κατά τη φάση εκπόνησης των έργων όσο και στην επιχειρησιακή φάση. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε ότι τα νέα μέσα από τα απλουστευμένα ε, και χαμηλότερου κόστου, είναι προσβάσιμα για όλες οι επιχειρήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να γίνεται αναφορά και στο ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών. Κάθε μήνα στην Ευρώπη εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρεοκοπούν διότι δεν τους εξοφλούνται τιμολόγια που έχουν εκδώσει έχουμε την οδηγία 7 του 2011 όσον αφορά τους όρους πληρωμής της εμπορικές συναλλαγές. Ε, αυτή η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους από τα κράτη-μέλη, διότι αυτές οι καθυστερήσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και για την υλοποίηση μιας πραγματικής ενίας αγοράς. Το θέμα δεν είναι να ελέγχουμε μόνο κατά πόσο οι πόροι έχουν όντω φτάσει στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι τα κονδύλια πηγαίνουν απευθεία και γρήγορα σε αυτέ, ότι φτάνουν σε αυτέ. Πρέπει να ελέγχουμε λοιπόν ότι οι δικαιούχοι είναι όντω απευθεία μικρομεσαίες επιχειρήσει. Οι διοικητικοί ικανότητε των τοπικών οργανισμών είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη ε, σύγχρονων επενδυτικών προγραμμάτων ε, και μακροχρόνιων που θα σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πρέπει επίσης με αυτή την έκθεση να προσπαθήσουμε μαζί με τους συναδέλφους να ασχοληθούμε με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικο-οικονομικές και ιστορικές μάλιστα πτυχές που για διάφορους λόγους σχετίζονται με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την πράσινη οικονομία θα ήθελα να αναφερθώ στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου ε, το 40% του κόστους της μεταπηδικής βιομηχανίας στην Ευρώπη ε, αποτελεί το... αποτελούν οι πρώτες ύλες ενώ το κόστος εργασίας είναι μόνο το 20%. Η βοήθεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βοηθήσει να επιτύχουμε αυτό το μηδενικό χιλιόμετρο που αναφέρουμε μέσω μιας οργάνωσης σε κλάστερ. Αυτή η τελευταία πτυχή θα ευνοήσει τοπικές επενδύσεις σε όλες τις περιοχές βάσει των παραδόσεων και των τοπικών τεχνογνωσιών. Ειδικότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικροεπιχειρήσεις, εκείνες δηλαδή με λιγότερους από 10 υπαλλήλου που αποτελούν σημαντικό ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεις και που μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίες καθημερινά όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις. Βάσει αυτή της πεποίθησης που δημιουργείται από την ανάγκη να γνωρίζουμε κατά πόσο εφαρμόστηκαν σωστά οι εργασίες μέχρι στιγμή, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμβάλλουν σε πραγματική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χάρη στην σωστή εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Θα ήταν λοιπόν εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή των συναδέλφων εισηγητών, σκιωδών εισηγητών και όλων των ομάδων που θα συμμετάσχουν. Θα δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα κατάλογο των επιχειρημάτων που, με τα οποία θα ασχοληθούμε βάσει του γενικού πλαισίου που σας παρουσίασα σήμερα. Σας ευχαριστώ και αναμένω τα σχολεία σας. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις. Πρώτα τους παρόντες. Ποιοι είναι παρόντες σκιώδεις. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Νταμάτο, για την εξαιρετική της έκθεση. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουμε 970 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης το ΦΕΝΤΕΡ. Από τη μία ε, θα έχουμε κονδύλια για οριζόντια στήριξη ε, για επιχειρηματίες σε διάφορους κλάδους και ε, σε νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς επίσης και κεφάλαια κινδύνου, δάνεια και εγγύησης δανείων, τα κλασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δημιουργούν δουλειές και βοηθούν να απέσει η ε, υπάρχουν και δημογραφικά προβλήματα και προκλήσεις. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και ταυτόχρονα να αυξήσει και το κατακεφαλήν ε, ΑΕΠ. Έτσι θα έχουμε ένα υγιή κλάδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία. Το 2013 έγινε μια ανάλυση που έδειξε ότι ε, η χρόνια υποχρηματοδότηση βλάπτει. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις τράπεζες, από τις χρηματαγορές ή από άλλες πηγές. Είναι πρόθυμες τώρα οι τράπεζες να αναλαμβάνουν κινδύνους σε τέτοιους καιρούς. Άρα 79% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ιδίους πόρους και έσοδα από τις δραστηριότητες τους που επανεπενδύουν τα κεφάλαια κινδύνου σχεδόν ανύπαρκτα στις μικρομεσαίες και Επίσης και το λεγόμενο δίκτυο Business Angels ε, που χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται επικελματική υποστήριξη ε, αυτών των ανθρώπων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν όμως την οικονομική δυνατότητα να έχουν ειδικέ υπηρεσίες ή να προσφεύγουν σε αυτές. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι υψηλής ποιότητας γιατί δεν έχουν τους πόρους για να καταφύγουν σε επαγγελματίες. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος. Χρειάζεται ειδικέ υπηρεσίες να παρέχονται ε, στις μικρομεσαίες με διαφορετικό τρόπο από τις μεγάλες. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε ένα περιβάλλον που να μπορούν να αναπτύσσονται και να ε, μεγαλώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και νέες δεξιότητες στην ψηφιακή αγορά. Έτσι, θα είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση, πιο σύντομες και πιο φθηνές οι διαδικασίες. Σε 19 κράτη-μέλη χρειάζονται τρεις μέρες για να ιδρυθεί μια εταιρεία, ενώ σε άλλες χώρες μπορεί να χρειάζεται από μία μέχρι πέντε μέρες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη 450.000 ε, εταιρείε ε, μεταφέρονται και δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι. Ο κύριος Οστρεβίτσιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για τους φιλελεύθερους θα ήθελα ε, και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Νταμάτα από το EFTD ε, για την έκθεση υλοποίηση ε, για λογαριασμό της Επιτροπής Ρέτζη. Πρέπει να επανεστιάσουμε την πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων ε στον αμφισβητή. Χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική για να επιτύχουμε τους στόχους μας και για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ε, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, είναι εξαιρετική η ευκαιρία που μα δίνεται με αυτή την έκθεση για έναν απολογισμό πεπραγμένο σε σχέση με την μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχή για να διπλασιάσουμε τις επενδύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να φτάσουμε τα 140 δις για την περίοδο 2014-2020. Ε, μία από ε, τι βασικέ μας πολιτικές προτεραιότητε, ε, ανέκαθεν και εξακολουθεί να είναι και τώρα, είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικής αποτελεσματικής ε, επιχειρηματικότητας ε, στην Ευρώπη και βελτίωση των συνθήκων ε, πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξανόμενες επενδύσεις, απλουστευμένοι κανόνες, εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα σε επιμέρους προγράμματα, διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μέσα τα χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της μεταρρυθμισμένης πολιτικής συνεχής της ΕΕ ναι, και Βασιζόμαστε στα διδάγματα που αντλήσαμε την προηγούμενη περίοδο, 2007-2013, όπου ε, υποστηρίξαν πάνω από 95 startup επιχειρήσεις και πάνω από 300.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα μέσα από αυτή την έκθεση για την εφαρμογή ε, των προγραμμάτων και τις βελτιώσεις που χρειαζόμαστε, τις απαραίτητες βελτιώσεις ούτως ώστε οι μικρομεσαίες ε, να μπορέσουν στο ε, έπακρο να υποφεληθούν από τις διαστατικές επενδύσεις και να εφαρμόσουν τις συστάσεις που προκύπτουν σε σχέση με τα εκρεμή προβλήματα. Κατά την σύνδεξη της έκθεσης θα πρέπει, συνάδελφοι, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να ε, αντικατοπίζουμε τις ε, απόψεις ε, των φορέων επιτόπου, διότι έχουν τις πιο ρεαλιστικές απόψεις και προσδοκίες και αυτό είναι στοιχείο κλειδί για μας, επειδή προσπαθούμε να βασιζόμαστε σε δεδομένα για να κατευθύνουμε την πολιτική συνοχή στο μέλλον. Συνάδελφοι, ελπίζω να είναι χρήσιμη η σημερινή ανταλλαγή απόψεων και να έχουμε σφαιρικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν με την υποβολή του τελικού σχεδίου έκθεση υλοποίησης. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτω συγγνώμη ε, για τη συνάδελφα που εξακολουθεί να μην είναι εδώ, αλλά παρόλα αυτά μου έχει στείλει τη θέση της. Η κυρία Κάλιτς ε, καλωσορίζει την πρωτοβουλία της κυρίας Νταμάτο συμφωνούμε με, μαζί της για τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με ε, την πρόθεση μιας εύρωστης οικονομίας ε, στις περιοχές των κρατών στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα ε, στα κονδύλια των διαφόρων ταμείων διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσουμε για την ευφυή εξειδίκευση, για την έρευνα και την καινοτομία να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να, γιατί αυτά θα είναι και η δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο μέλλον θα, οποιασδήποτε πληροφορίε λάβει η κυρία Νταμάτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ε, έκθεση πραγμένων για τι ε, ε, συνέργειε των διαφόρων ταμείων για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα ήταν καλό να τι μοιραστεί μαζί μα. Θα θέλαμε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα στην τελική έκθεση. Ε, και προσβλέπουμε και ε, στη μελλοντική συνεργασία με την εισηγήτρια κυρία Νταμάτο. Σας ευχαριστούμε. Πανίστε, Ρόι ε. και Μπρέσο. Ευχαριστώ Ο κύριος Σίκου που είναι σκιώδης εισηγητής μας και συμπατριώτης σας κυρία Νταμάτο μου δώσε μερικά σημεία να τα πω εγώ σύντομα. Έχετε δίκιο. Στην αρχή μιλήσατε για την ανταγωνιστικότητα. Ε, περί αυτού πρόκειται. Και από εκεί ξεκίνησε και η ε, πρωτοβουλία μας. Ε, Βεβαίω η χρηματοδότηση είναι σημαντική, αλλά ο τελικός στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να δούμε ότι τα ταμεία μας είναι ένας κρίκος στη μεγαλύτερη αλυσίδα και εκεί θα πρέπει να αναζητούμε συνέργειες. Δηλαδή, εμείς έχουμε περιορισμένες δυνατότητες, αλλά συμπληρωματικά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα μέσα και εργαλεία στην αγορά για να βοηθήσουν. Κοιτάξτε το εύση το Τραμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων, 75 ε, δισεκατομμύρια ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ε, να συνεργάζονται και τα διάφορα ταμεία μεταξύ τους και το λέει και ο εισηγητής μας ο Σκιώδης. Τρίτον, συνεργασία διασυνοριακή και διεθνής. Κοιτάξτε ένα τομέα ας πούμε όπως είναι το διαδίκτυο, η ψηφιοποίηση. Είναι τεράστια η αγορά που διανοίγεται Εάν φύγετε όμως από τα αστικά κέντρα και φτάσετε στην Ήπεθρο, τι να το κάνετε αν δεν έχετε τις συνδέσεις, όσο καλές ε, ε, δυνατότητες και να έχετε. Η Επίτροπος Βιανκόφσκα ε, παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες την πρότασή της για τις νεοφύης επιχειρήσεις και τις υπόλοιπες που δεν έχουν πρόσβαση Άρα χρειάζεται πάρα πολύ ε, μεγάλη ε, συνεργασία. Το ξέρω ότι και εσάς θα απασχολεί αυτό. Το συζητήσαμε και στην προηγούμενη, στην εδαφική συνεργασία, στο προηγούμενο θέμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε για τις εκθέσεις για το άρθρο 13, 16, συγγνώμη, γιατί το 3 είναι θεματική συγκέντρωση. Και ε, περιμένουμε αποτελέσματα. Όταν κάνεις εκθέσεις εκτέλεσης και εφαρμογής πρέπει να κοιτάς αριθμητικά στοιχεία για τα αποτελέσματα γιατί εκεί μετράς εάν έχουν ε, ε, αποδώσει οι πολιτικές σου. Εγώ περιμένω πάρα πολλά τέτοια αριθμητικά στοιχεία στις εκθέσεις. Μπορείτε και εσείς να το συμπεριλάβετε στη δική σας έκθεση. Τι άλλο να σας πω. Στη ΣΤΟΑ ήμουν σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση που ξέρετε ότι είναι η μονάδα ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον Πάουλ Ρούμπιχ και άλλους ιδιαίτερα από τον κύκλο της Επιτροπής Ήτρε και λέμε τι γίνεται εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε ένα χάρτη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε ένα σωρό νέα εργαλεία με κεφάλαια κινδύνου. Υπάρχουν δυνατότητε στήριξη για νεοφυεί επιχειρήσει. Έχουμε πολλά πράγματα για τι μικρομεσαίε. Όλα αυτά όμω συνδυάζονται μεταξύ τους. Και ήταν διάφοροι εμπειρογνώμονες που μίλησαν και εντός και εκτός κοινοβουλίου και κανείς δεν αναφέρθηκε στη δική μας επιτροπή και στην πολιτική συνοχής. Μα εμείς δεν έχουμε ρόλο εκεί να διαδραματίσουμε αλίμον θα πρέπει να υπάρξει παράγραφος και χωριστή για το τι γίνεται με τα μέσα που έχουμε για την περιφερειακή πολιτική και πώς μπορούν αυτά να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά θα πρέπει να μπουν στην έκθεση. Ο καθένας να κοιτάει τις δικές του βέβαια επιδόσεις, αλλά και πώς μπορεί να συνεργάζεται. Α, και ένα τελευταίο που ξέχασα. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στις προσπάθειες που καταβάλει το κοινό ερευνητικό κέντρο στη Σεβίλη. Στο τέλος της εβδομάδας θα μεταβούμε εκεί με αντιπροσωπεία και ε, υπάρχει ένα ε, θέμα που λέγεται ε, entrepreneurial discovery, δηλαδή ανακαλύπτουμε ε, στις επιχειρήσεις, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στην ε, πληροφορική, στο τέταρτο στόχο για το περιβάλλον, ε, όλη η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και με την εξειδίκευση, αλλά το πώς θα γίνει συγκεκριμένα αυτό πράξη είναι πάρα πολύ ουσιώδης και ε, αξίζει προσοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Μπρέσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, και ο δικός μας ε, και ο ο Ανδρέα Κοτσολίνο έχει κολλήσει στην κίνηση των Βρυξελών. Θα κάνω λοιπόν εγώ στη θέση του κάποια παρατήρηση, κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεση αυτή που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και να ευχαριστήσω την κυρία Συγγετρία ε, που μας πρότεινε ένα θέμα σαν αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι παρότι αυτή η πολιτική είναι μια κλασική πολιτική της πολιτικής συνοχής, η υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω λοιπόν παρόλα αυτά ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που στο πλαίσιο του νέας προγραμματικής περίοδου παρεμβαίνουμε σε ένα παραγωγικό ιστό που πλήττεται από την κρίση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέφεραν ιδιαίτερα κατά το διάστημα της κρίσης. Έτσι λοιπόν τα μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή ε, ενεργοποιούνται είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβουμε κατά πόσο η παρέμβαση αυτή μετά την κρίση ε, αν έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα μέσα ειδικότερα όσον αφορά το γεγονός ότι από την κρίση βγαίνει κανείς με περισσότερες καινοτομίες Τι γίνεται λοιπόν με την έρευνα, με τη συλλογική ανάπτυξη της έρευνας, γιατί συχνά μιλάμε για επιχειρήσεις πολύ μικρές. Τι ακριβώς υλοποιείται λοιπόν ε, συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων τύπου κλάστερ, ομάδες, όμιλοι, κοινά ερευνητικά προγράμματα που, στα οποία συμμετέχουν πολλοί διάφοροι ενδιαφερόμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κέντρα ε, ε, εφαρμοσμένων ερευνών κτλ. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη, είναι πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική η μεταφορά τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεπώς, ε, πόσα προγράμματα υπάρχουν ε, και πώς έχουν δομηθεί αυτά. Υπάρχουν, ε, είναι καλοφτιαγμένα λοιπά Τρίτο θέμα, ε, τρίτο θέμα που πολλοί συνάδελφοι μάλιστα ανέφεραν, αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν ιδιαίτερα από τα οικονομικά προβλήματα, δηλαδή το κόστος, τις δυσκολίες εξέβρεσης κονδυλίων Ακόμα και τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Ε, χαμηλότερα από το 0, αλλά αυτά τα επιτόκια δεν διαφέρουν στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε τι χρηματοοικονομικά μέσα υπάρχουν ε, και καινοτόμα μάλιστα θεματικά επενδυτικά ταμεία τι υπάρχει ε, που να προσαρμόζεται ε, στα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να τις βοηθήσουν, να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό το γέριο παράγοντα που θα τις βοηθήσει να βγουν από την κρίση, όχι μόνο με την καινοτομία. Ε, από την, θα βγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κρίση με την καινοτομία, αλλά η καινοτομία κοστίζει. Ε, πώς χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε εποχές τέτοιες πολύ χαμηλού κόστους του χρήματος. Ε, τώρα, αν δεν μπορούσε η συγγήτρια με τη βοήθεια της Κομισιόν να μας ε, περιγράψει το πλαίσιο βάσει του οποίου οι αρχές προγραμματισμού έχουν και να και ενισχύσει την υποστήριξή τους προς τις μικρόμεσες επιχειρήσεις για να βγουν αυτές από την κρίση. Ε, αν θα μπορούσε λοιπόν να μας περιγράψει αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς η πολιτική συνοχής πώς η πολιτική συνοχής ε, καταφέρνει να βοηθήσει ε, τις μικρόμεσες επιχειρήσεις να βγουν από την κρίση ε, ίσως ε, και πριν ε, τελειώσουμε όλες τε, τα σχόλια να έρθει βέβαια, να βρίσκεται εδώ ο και ο συζητητής, αλλά προς το παρόν δυστυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much, but we have... Uh, Σας ευχαριστούμε. Δεν πειράζει. Γνωρίζουμε τη θέση του. Για να δούμε τώρα αν ε, ο εκπρόσωπος Επιτροπής θέλει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μας δίνετε την ευκαιρία για, αυτή το, για αυτό το θεματικό στόχο 3 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να κάνουμε και εμείς κάποια σχόλια. Όταν αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, τους δείχναμε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι ένας ε, γνώμονας, ε, μπορούσαν να ακολουθήσουν για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και περιοριζόμαστε σε αυτά που λέει ο κανονισμός. Startups, ε, νέες εταιρείες, ε, διεθνοποίηση, ικανότητα, μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό για τις επιχειρήσεις, ε, ενθάρρυνση της καινοτομίας και αυτό Τόσο θεματικός στόχος 3 ε, δεν τελούσε υπό την αίρεση της ε, εφίους ε, εξειδίκευσης, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε την εφή εξειδίκευση ως εξάντε προϋπόθεση στο θεματικό στόχο 1. Στο 3 όμως δεν υπήρχε αυτή η αίρεση, οπότε τα κράτη-μέλη σε κάποιες περιοχές διοχέτουν διοχέτευαν ε, τα κονδύλια στον στόχο 3 γιατί ε, τον ε, κλάμεραν ως ευκολότερο. Διότι έχουμε και το Small Business Act σε σχέση με το πρώτο στόχο, αυτό συνεχίζεται και να σας θυμίσω περί πρόκειται, είναι η ταχύτητα ίδρυσης, στην ίδρυση των επιχειρήσεων, η παρακολούθηση εφαρμογής του Small Business Act, και τα προβλήματα επίσης ήταν και καθυστερήσεις στις πληρωμές. Την εξάντερεσιμότητα την είχαμε ούτω ώστε ε, να παίρνουν στα σοβαρά ε, τους ε, κανόνες τα κράτη-μέλη και άρα σε αυτό το θεματικό στόχο 3 δεν είχαμε θέματα με καθυστερήσεις πληρωμών. Σε κάποια κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις ασκήθηκε πίεση για να πάνε τα κονδύλια στον πρώτο θεματικό στόχο, ε, ούτως ώστε να ανέβουμε σε σχέση με την αλυσίδα αξίας. Η τάση σε ορισμένα κράτη-μέλη ήταν να μην διατηρηθεί η κατάσταση, αλλά να μεταφερθούν τα κονδύλια και να μπουν στην, στον τρίτο θεματικό στόχο. Βλέπετε και στα στατιστικά στοιχεία ότι μεγάλωνε διαρκώ το μερίδιο. Δηλαδή, όλα είναι και περισσότεροι όλα τα κονδύλια από τον πρώτο στόχο πηγαίναν στον τρίτο. Παρόλα αυτά, γιατί υπάρχουν και επιπτώσεις, υπάρχουν τομείς παρέμβασης και οι γενικές επενδύσεις είναι ο πιο σημαντικός. Αυτό σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Στο θεματικό στόχο 3 μπορούν οι επιχειρηματίες να έχουν ολόκληρο το φάσμα των επενδύσεων, να τις έχουν δηλαδή ως επιλέξιμες. μέσα από τα επιμέρους μέτρα. Το ένα, που είναι, το ένα στοιχείο που είναι θετικό είναι ότι ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα νέα οικονομικά μέσα. 10 δις στον τρίτο στόχο θα ε, σχετίζεται με τα νέα οικονομικά μέσα. Οτιδήποτε σχετίζεται με τις γενικές επενδύσεις θα υποστηρίζεται από ε, δάνεια, από εγγυήσεις, ό,τι έχει σχέση με νέα χρηματοδοτικά μέσα δηλαδή. Για τις ε, συνέργειες θα ήθελα να πω πως με τη στρατηγική 2020 έχουμε το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, έχουμε ε, το θέμα αριστείας, δηλαδή τι γίνεται στα πλαίσια του 2020 κάποια προγράμματα που δεν λάμβαναν χρηματοδότηση, όχι επειδή δεν ήταν καλά, αλλά γιατί στον ορίζοντα 2020 δεν υπήρχαν άλλα κονδύλια, μπορούν τα κράτη-μέλη περιοχές να χρησιμοποιήσουν τώρα αυτά τα προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα, στο μέτρο που όμω συνάδουν και με τη διαδικασία τη ευφυού εξειδίκευση. Για την ε, απλοποίηση, γιατί είναι βασική μέρημνα τη Επιτρόπου μα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία με ομάδε εργασία και ε, υπάρχει υποστήριξη του streamlining για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος πάντων, όταν εσείς αναφέρατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να βοηθήσει την εισηγήτρια για να δούμε τις καινοτόμες προσεγγίσεις των κράτων μελών και των περιοχών σε σχέση με ε, τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα σας έλεγα ότι χωρίς να προσπαθούμε εμείς να ε, βρίσκουμε fast track διαδικασίες για να βρούμε νέα κονδύλια, γιατί υπάρχουν και οι κανόνες και εξακολουθούν να ισχύουν, υπάρχει παρόλα αυτά περιθέριο σε επίπεδο κρατών μελών και περιοχών για streamlining των διαδικασιών χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ανταμάτο, θα θέλατε να απαντήσετε ή να μας παρουσιάσετε κάποια συμπεράσματα. Να ευχαριστήσω όσους ε, μίλησαν Ακούσαμε νέες ιδέες, ε, νέα αιτήματα για να εμβαθύνουμε κάποια θέματα από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. Θα τα λάβουμε όλα υπόψη και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε μια επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Can move to the... Και τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Πού είναι? Μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, είναι ε, προς την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Υπολογισμού. Η συγκήτριά μας είναι η κυρία Ιβάνα Μάλετιτς, είναι απαλλαγή 2014 Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού δηλαδή. Ποιο θέλει, ε, ο κύριος Μανίστεροι. Ροϊ. Ε, να αυτοσχεδιάσω λίγο τώρα εγώ, γιατί γενικά σήμερα απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Ε, δεν ήταν γραφτό, δεν τα κατάφεραν οι δικοί μας να έρθουν. Έχω κείμενο και μπορώ και να σας το διαβάσω γρήγορα. Είναι και στα αγγλικά. Λοιπόν, το διαβάζω αγγλικά. Πάμε. Αξιότιμα μέλη το ελεκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεση το 2014 σημείωσε ότι έχουμε 4,4% ε, ποσοστό σφαλμάτων στις πληρωμές. Υπάρχει μια μικρή μειωσή σε σχέση με την περσινή ετήσια έκθεση που ήταν 4,3%. Μια μικρή αύξηση. Πάντως εκεί κάπου ε, κινειται 3,4 από 4,3-4,4 αλλά γενικότερα είναι υψηλότερο από το 2% που θεωρείται αποδεκτό σφάλμα. Επιπλέον ε, η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο αντίστοιχο τίτλος, ε, ε, βλέπει τα ασφάλματα να μειώνονται σε σχέση με την περσινή πάλι έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. 5 0,7% ε, είναι τα σφάλματα για το 2014, ενώ το 2013 ήταν 5,3%. Τα υψηλά επίπεδα σφαλμάτων και οι ατασταλίες και οι παρατυπίες υπονομεύουν την επενδυτική εμπροκειμένου ε, ε, την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις όλο αυτό στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φαίνεται και από άλλη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου δηλώνουν ότι παρόλο που οι απάτες έχουν μειωθεί στην πολιτική συνοχής, υπάρχει αρνητικός ε, χρηματοδοτικός αντίκτυπος ε, μεγαλύτερος κατά 76% σε σύγκριση με το έτος 2013. Σε περίπτωση ε, σφαλμάτων που δεν είναι απάτες, αν είναι παρατυπίες και τα λοιπά, αυτά αυξήθηκαν και σε σύγκριση με το 2013. Το αποτέλεσμα αυτό απορρέει από το γεγονός ότι είναι ανεπαρκής η έλεγχη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών φυσικά. Και καθώς επίσης ε, δεν είναι καλή και χρηστή η οικονομική διαχείριση. Γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές παρατυπίες. Και εδώ είναι το σημαντικό και το τονίζω. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκες οι διαδικασίες. Οι κανονισμοί και οι κανόνες και τα λοιπά ε, προκαλούν ε, δυσκολίες στους τελικούς χρήστες και δικαιούχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν πει και ε, στο παρελθόν ότι βελτιώνουν τους μηχανισμούς για τους ελέγχους, για τη διαχείριση και τα λοιπά οικονομικά. Επιπλέον, η ενημέρωση που θα ήταν πολύτιμη για την πρόληψη αυτών των απατών δεν χρησιμοποιείται και δεν αξιοποιείται πλήρως. Άρα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο ενεργά στην ανταλλαγή γνώσεων ε, ε, και βελτίστων ε, πρακτικών για να μειωθεί ο ο αριθμός και το ποσοστό σφαλμάτων και παρατυπιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει για να απλοποιηθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες, διατηρώντας όμως σε κανονικό επίπεδο στην οικονομική διαχείριση με στόχο πάντα την επιθυμητή ισορροπία για τους τελικούς δικαιούχους. Να μην σταματάνε πληρωμές, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαπιστώνονται κάποιες παρατυπίες ή σφάλματα που δεν είναι απάτες. Να μην σταματάει η χρηματοδότηση, διότι αυτό θα κάνει τα έργα να κινδυνεύουν. Σε περίπτωση που είναι απάτες, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εφαρμόσει τους αντίστοιχους κανόνες. Συμπέρασμα. Θα πρέπει δαπάνες να είναι προσανατολισμένες περισσότερο στο αποτέλεσμα και αυτό έχει να κάνει και με τις συμφωνίες των κρατών μελών και τα συμβόλαια και δημιουργεί ε, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες και μια πιο υπεύθυνη διαχείριση ε, των χρημάτων των φορολογουμένων. Αυτό το κείμενο θα σας το δώσω για τα πρακτικά, γιατί είναι του εισηγητού και θα δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Και σε εσά εναπόκειται τώρα να μου πείτε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τώρα κάποιους τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, κύριε Βόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ήταν εδώ εισηγητής θα τον ευχαριστώ και εγώ για τις προτάσεις του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εισηγητής ο κ. Λάμπερτ ε, ανέφερε ότι παρατηρείται χαμηλή μείωση του ποσοστού σφάλματος ε, για την ευρήματα της ε, πολιτικής συνοχής και για το γεγονό ότι το σφάλμα δεν είναι το ίδιο με την απάτη. Ξέρετε, ορισμένοι φορές σε άλλες επιτροπές επίτηδες θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα, ενώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Χαίρομαι επίσης που στις προτάσεις τη εισηγήτρια επισημαίνεται ο σημαντικό ρόλο των κρατών μελών ε, στη μείωση του ποσοστού σφάλματο. Γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα σφάλματα ουσιαστικά τα διαχειριζόνται τα κράτη-μέλη. Ένα πράγμα που δεν περιλαμβάνεται στη στάση, αλλά πιστεύω θα έπρεπε να αναφέρεται, θα ήταν το γεγονό ότι σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανείχνευση των μη διορθωμένων σφαλμάτων. Οπότε τα κρατη έχουν μεγάλη ευθύνη. Θα μπορούσε να αναφερθεί αυτό μέσω κάποιε τροπολογίε ενδεχομένω. Κάτι άλλο σημαντικό που αναφέρει ο εισηγητής είναι η απλούστευση. Σε κάθε επίσκεψη, είτε της Επιτροπής Ρέτζη, είτε της Επιτροπής Ελεκτών Προπολογισμών, ε, όπου και να πηγαίνουμε, πάντα μας λένε το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει για να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων είναι το να υπάρξει ακόμη περισσότερη απλούστευση και το λέμε όπου πάμε. Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα όπου ένα σύνολο κανονισμών ε, καλύπτουν τους πέντε βασικούς τομείς, η δυνατότητα εφάπαξα πληρωμών, ε, συνεργειών μεταξύ διαφορών ταμείων, όλα αυτά βελτιώνουν την κατάσταση. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέλλον για να προσθέσουμε ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Ε, κάποιου είδους κοινοί κανόνες. Ε, να δούμε και τους κανόνες ε, των δημοσίων προμηθειών, διότι ξέρετε το 50% των σφαλμάτων που βρίσκει το ελεκτικό συνέδριο αφορά ζητήματα δημοσίων προμηθειών, οπότε μπορεί να γίνει κάτι εκεί πέρα, ίσως για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον. Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν στο μέλλον για να προσθεθούν ακόμη περισσότερα τα πράγματα για τα κράτη-μέλη, για τους δικαιούχους, για τις περιφέρειες, για τους ελεκτές επίσης. Ε, Βελτιώντα λοιπόν, ε, απλουστεύοντα ακόμη περισσότερα τα πράγματα, πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενη και είμαι εγώ. Οπότε θα συνεχίσω με τις ρεξικέλευτες αυτές διαδικασίες που είπαμε και ναι ξέρω. Ναι θα σα δώσω το λόγο σε εσά, κυρία Ταμαντζήτς. Ναι, εντάξει. Λοιπόν αγαπητοί συναδέλφοι Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία απαλλαγή αποτελεί σημαντικό βήμα στις δυνατότητες εξέταση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Στην Επιτροπή Ρέτζη αποτελεί ευκαιρία προβληματισμού να δούμε ποια υπήρξαν τα κυριότερα επιτέγματα όσον αφορά την εκτέλεση του ετήσιου προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική συνοχή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την συγγήτρια, συγγνώμη τον εισηγητή, την εισηγήτρια την κυρία Εύανα Μελέτητς από την ομάδα ΕΛΚΑ για την γνωμοδότησή της ε, Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΡΕΤΖΙ καθώς και την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2014 η, την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το 2014 και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα θα ήθελα να επιστήσω ε, την προσοχή σας στα ακολουθά θέματα. Το 2014 η πολιτική συνοχή, όπως και τα περασμένα έτη, θεωρήθηκε από το ελεκτικό συνεδριό ως τομέας πολιτικής ε, ιδιαίτερα επιρρεπής σε σφάλματα. 5,5 ήταν το ποσοστό σφάλματων, χωρίς μεγάλη διαφορά μεταξύ σφάλματων δημόσιες ε, προμήθειες, καθώς και επιλεξιμότητα είναι οι τομείς όπου παρατηρούνται τα περισσότερα σφάλματα. Από αυτή την έψη, λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω τα εξή. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιμαστούν πάνω απ' όλα στην σχεδιασμό κατάλληλων προληπτικών μέτρων, έγκαιρη πληροφόρηση και αποτελεσματική εκπαίδευση και καθοδήγηση προ τι εθνικέ αρχέ για του ε, εντοπισμένου κινδύνου, απλούστευση των διαδικασιών διαχείριση και ελέγχου στα προγράμματα και στην υλοποίησή του ώστε να αποφεύγονται σφάλματα και το αυξημένο επίπεδο διακοπών εργασιών και πληρωμών. Η αποτελεσματική εκπαίδευση και η καθοδήγηση προς εθνικές αρχές ε, σε σχέση με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, ειδικότερα όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες ε, και τους κανόνες ε, κρατικών ενισχύσεων, είναι σημαντικές πτυχές για την πρόληψη των σφαλμάτων. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν να υλοποιήσουν στοχευμένα και έγκαιρα και επίκαιρα μέτρα γρήγορα μέτρα για να ενισχυθούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική αυτή. Επειδή οι δημοσίες προμήθειες είναι ένας τομέας με πολλές ε, αρνομιομορφίες, καλωσορίζω το νέο κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΥΦ 2014-2020 με την εξαντιορισμότητα όσον αφορά τη τις δημόσιες προμήθειες. Είναι απαραίτητο για τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν πληρούν την εκ των υστέρων αιρεσιμότητα να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν τα συμφωνημένα σχέδια δράση μέχρι το τέλος του 2016. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενσωματώσουν και να μεταφέρουν γρήγορα το πακέτο του 2014 των οδηγιών δημοσίων προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους νομοθεσία μέχρι την 18 Απριλίου του 2016. Ταυτόχρονα η Κομισιόν θα επιτηρεί αυστηρά τη διαδικασία αυτή παρέχοντας την απαραίτητη καθοδήγηση και τεχνική αρρωγή προς τα κράτη-μέλη για τη σωστή μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Συμφωνώ λοιπόν πλήρως με τους υπόλοιπους και Θα πρέπει να ε, δούμε πώς μπορούμε να απλωστεύσουμε περισσότερα τα πράγματα, να προσφέρουμε καλή καθοδήγηση και ενημέρωση στις ε, αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο σφαλμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μάλτες για την έκθεση και για τις προτάσεις που κάνει. Με τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες των κρατών μελών και την ανεπάρκεια των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η καλή διαχείριση και η ε, μέγιστη αξιοποίηση των κονδυλίων. Πολλές φορές ε, δεν υπάρχει γνώση των κανόνων, των περίπλοκων κανονισμών και σε αυτό μπορούν να αποδοθούν πολλά λάθη. Έτσι, με απλούστευση των κανόνων, πολλές παρατυπίες που δεν συνιστούν απάτη θα ε, μειωθούν ως προς τον αριθμό. Η ε, ομάδα υψηλό επίπεδο ανεξαρτήνων εμπρογνωμών για την επόπτωση και την απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιώχους των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη νομοθεσία έχουμε στη διάθεσή μας πλέον αποτελεσματικά μέσα. Όμως χρειαζόμαστε και μια καλή συμφωνία Προτού εκδώσουμε συστάσεις, διότι απλούστευση σε ένα κράτος μπορεί να οδηγήσει σε περιπλοκότητες, ε, σε πιο περίπλοκες διαδικασίες σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, το βασική μας μέρημα θα πρέπει να είναι η μείωση του διοικητικού άχθους για τους δικαιούχους και θα πρέπει η επόπτευση να βασίζεται σε αποτελέσματα των προγραμμάτων με το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου. Ε, και κύριε Βάνο, πάλι και εσείς εκπροσωπείτε την σκιώδης γιατριά Ναι, ζητώ συγγνώμη από πλευρά τη. Ε, και θα ήθελα να σας διαβάσω τη θέση της. Ε, το 2014 είναι η πρώτο έτος υλοποίησης ε, του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και του νέου πλαισίου από το 2018 έως 20. Είναι πολύ μικρό μερίδιο των κονδυλίων 2014 που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη για τα προγράμματα νέας γενιάς. Μιλάμε για την νέα περίοδο 2014-2020, για την περίοδο συνοχής υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις και σημαντικά κολλήματα που δεν μας επέτρεψαν ομαλώς να μεταβούμε στη νέα προγραμματική περίοδο και να συνεχιστεί η οικονομική ροή και χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Μετά τι καθυστερήσει, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τι ε, συνέπειε τη καθυστέρηση ω προ την υλοποίηση των προγραμμάτων και να αντλήσει τα δέοντα συμπεράσματα. Επιπλέον, παρά την ανάγκη διαπίσπευση τη υλοποίηση των προγραμμάτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην ποιότητα των προγραμμάτων για να μην τη θυσιάσουμε για να επισφέσουμε τη διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί η καταπολέμηση της απάντησης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε επίσης να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, ε, ούτως ώστε να αρχίσουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank, you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, ζητώ συγγνώμη, κάποιον ξέχασα. Okay. The floor is yours. Thank you. Όχι, εντάξει, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις προτάσεις. Θα τις διαβιβάσω και στην Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την απαλλαγή 2014. Έχουμε τέσσερα μικρά σχόλια εμείς για τις προτάσεις αυτές. Πρώτον, γιατί πρώτη πρόταση η υπόδειξή σας ε, που έχει να κάνει με την αύξηση των σφαλμάτων ή το ποσοστό των αντιστοιχών. Κοιτάξτε ε, με προσοχή την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου θα δείτε αλλού αύξηση και αλλού μείωση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. methods uh, Γιατί ε, διαφέρει η μεθοδολογία καταμέτρησης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, έχει σταθεροποιηθεί το ποσοστό των ε, σφαλμάτων στην πολιτική συνοχή και κυμαίνεται στο 5 με 7% για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έκτοτε μειώθηκε, αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα σημερινά, με το 2014. αλλά παραμένει αρκετά υψηλό και έχει μειωθεί και σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006. Ανέφερε κάποιο μέλος της Επιτροπής σας ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι παραστάτε στα κράτη-μέλη, στο πλευρό μας, για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα σφάλματα. Το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει ότι 40% των ποσοτικοποιημένων σφαλμάτων που έχουμε μετρήσει δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ε, από τις εθνικές αρχές και θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί μάλλον, να το είχαν βρει τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, Χαιρόμαστε που κάνετε διάξη ανάμεσα στις παρατυπίες που δεν συνιστούν απάτη και τις απάτες. Καλό είναι αυτό. Τρίτον. Απλούστευση. Αυτό είναι και το σύνθημα της Επιτρόπου Κρέτσου. Υπάρχει πραγματικά αντίστοιχη ομάδα υψηλού επίπεδου που έχει συσταθεί για να απλοποιήσει τις διαδικασίες και τα συστήματα και αυτό ενδιαφέρει πολύ την κυρία Κρέτσου. And the, the fourth... Ε, και το τέταρτο που είπατε ήταν η εστίαση στα αποτελέσματα. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εστίαση στα αποτελέσματα, δηλαδή δεν είναι προσανατολισμένο και σχεδιασμένο το πρόγραμμα έτσι, ε, ώστε να στρέφεται προς τα αποτελέσματα. Από πού το συνάγουν αυτό, είναι κάπως ε, πρόεμο το στάδιο για να προχωρούν σε τέτοια προθύστερα συμπεράσματα. Τη 17 Δεκεμβρίου στην Ακρόαση, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και για την έκθεση τη λεγόμενη του άρθρου 16 που γύρω στις 15 Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί και θα λάβει γνώση και το Κοινοβούλιο όλων αυτών των θεμάτων και με ποιον τρόπο λειτουργεί το νέο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στραμμένο σε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Άλλα ε, συμπερασματικά σχόλια εξ ονόματος της εισηγήτριας, κύριε Βανίστερο, ε, ε, δεν μπορείτε προφανώ, Τι να κάνω, έχω σημειώσει με μεγάλη επιμέλεια και θα τα διαβιβάσω αρμοδίως και θα τα συμπεριλάβει με βεβαίως στην γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την γνωμοδότηση αυτή Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και πάλι είναι η ίδια με την προηγούμενη έκθεση. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο που φτάσαμε έχουμε εξαντλήσει τη σημερινή μας ημερήσια διάταξη και θα συνεχίσουμε και κλεισμένο, μάλλον στη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Να παραμείνουν οι συντονιστές. Άντε. Κάντε ένα κουράγιο ακόμα. Τελευταίο.